Bonjour tout le monde. Nous commençons notre réunion par l'adoption de l'ordre. Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Ξεκινήσουμε με την έγκριση τη εμερήσια διάταξη. Επειδή ο κύριο Ντέβα δεν θα είναι εδώ στο τέλο ε, τη μέρα, στο σημείο 13 θα το εξετάσουμε για την Ελία, θα το εξετάσουμε αύριο το πρωί μετά το σημείο 27. Το σημείο δηλαδή του κύριου Ντέβα, πρωτόκολλο Συμφωνία Ελευτική Σύμπραξη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ομόσπονδων Πολιτειών Μικρονησία, θα είναι αύριο το πρωί. Ε, εγκρίνεται η μέρη σε διάταξη. Ωραία. Τώρα, έχετε πάρει τα πρακτικά των συνεδριάσεων 25ης και 26ης Οκτωβρίου, όπως επίσης 8ης και 9ης Νοεμβρίου και 9ης Δεκεμβρίου. Αν έχετε παρατηρήσεις, να το πείτε στη γραμματεία παρακαλώ πριν από το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης. Εφόσον δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, τα πρακτικά αυτά θεωρούνται εγκεκριμένα. Τώρα, για τα πρόσφατα γεγονότα, έχω να κάνω κάποιες, κάποια σχόλια. Η Τινησία δεν είναι βασικά δικιά μας αρμοδιότητα, Ήθελα όμως να μιλήσω λιγάκι για το κίνημα ιστορικής απελευθέρωσης που είχαμε στην χώρα και έχουμε στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Οι οικονομικές εξελίξεις και η οικονομική κατάσταση σίγουρα είναι ένα βασικό στοιχείο για την αξιοπρέπεια των λαών. Δεν φτάνει όμως, ιδιαίτερα όταν ε, δεν επωφελείται από την οικονομική κατάσταση παρά μόνο μία μικρή ελίτ ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χρηστή διακυβέρνηση αποτελούν αξίες αναγκαίες και απαραίτητες αναγκαίες για τους λαούς. Οι αξίες αυτές είναι και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν πρέπει να τις υπενθυμίζουμε συνεχώς και να στηρίζουμε τους λαούς οι οποίοι επιθυμούν να χαίρουν των αξιών αυτών και να φροντίζουν για τη δημοκρατία που διαθέτουμε. Για την Τινησία λοιπόν για μένα είναι πολύ βασικό, αλλά και για όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, να στηρίξουμε με όλη μας τη δύναμη τις διαδικασίες των δημοκρατικών αυτών αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο τώρα για τις δικές της ανακοινώσεις. Ο κύριος Ντομίνικο Ρώσα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω μερικές πληροφορίες να σας δώσω τώρα στην αρχή του 2011. Ξέρετε ότι από 1η Ιανουαρίου έχουμε τη συγχώνευση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της ε, ΕΚΟ. Σε αυτό το στάδιο είμαστε σε μεταβατική περίοδο, όπου έχουμε ένα οργανόγραμμα το οποίο αποτελεί συνοθήλευμα των δύο γενικών ε, διευθύνσεων. Προσπαθούμε όμως να το κοιτάξουμε πιο προσεκτικά και να δούμε πώς θα έχει το νέο οργανόγραμμα, το οποίο θα αντικατοπτρίζει από τη μια μεριά τις πολιτικές προτεραιότητές μας και από την άλλη μεριά θα δίνει μεγαλύτερη σημασία στην δράση της γενικής αυτής διεύθυνσης της νέας έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ανάπτυξη. Σίγουρα έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Ξέρετε ότι κάποιες ε, ε, ενότητες, κάποιες ε, υπηρεσίες επικαλύπτονται αυτή τη στιγμή και πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο να δουλέψουμε. Πιστεύω ότι πάντως ότι με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε σε αυτό που έχει ζητήσει κατά το παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή μεγαλύτερο ορθολογισμό τις δράσεις μας και τις δράσεις των διαφόρων φορέων που συνεργάζονται στα πλαίσια της συνεργασίας. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα έχουμε ολοκληρώσει επίσης την πρωτοβουλία για τους στόχους της χιλιετίας. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει ανακοίνωση στις χώρες ΑΚΕ για το πώς η πρωτοβουλία αυτή που είναι επιπλέον στήριξη για να επιτεθούν οι στόχοι της χιλιετίας από τη μια και από την άλλη έχουμε και τα αποτελέσματα του δεύτερου ΦΕΔ στα μέσα της διαδρομής, όλα αυτά θα είναι έτοιμα. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω για το ότι προς το παρόν έχουμε ένα τύπο Συμβούλιο Ανάπτυξης που καθορίστηκε από την Ουγγρική Προεδρία και από την είπατε εκπρόσωπο για τις 22 Φεβρουαρίου. Συνήθως οι Πρόεδρός σας και ο κύριος Μισελ ε, ως ε, ε, συμπρόεδρος της Γενικής Διεύθυνσης συμμετέχουν. Η Επιτροπή πάντως προσπαθεί να δει ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διάσκεψη για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη αρχές Μαΐου του 2011. Αυτά είχα να πω και από εκεί και πέρα ευχαρίστως να σας απαντήσω αν έχετε ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η έκθεση δεύτερη ανάγνωση Τώρα για τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Έχουμε δύο νομοθετικά ε, θέματα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Ε, συστάσει σε δεύτερη ανάγνωση που είναι η αναθεώρηση στα μέσα της διαδρομής του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και υπάρχουν και τα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα. Ε, σε πρώτη ανάγνωση 10 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του για τις δύο αυτές υποθέσεις. Και σύμφωνα με τον κανονισμό, οι δύο αυτές υποθέσεις προσθέθηκαν στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας για σήμερα. Κανονικά, τυπικά, πρέπει να επιβεβαιώσουμε τον εισηγητή μας για τη δεύτερη ανάγνωση. Συμφωνείτε με τη σύσταση των συντονιστών να επιβεβαιώσουμε ως εισηγητή από τη μια τον κύριο Μίτσελ για την αναθεώρηση του μέσου συνεργασία για την ανάπτυξη για την άλλη μεριά του κ. Γκέρεν για τα νοθευτικά μέτρα για την μπανάνα. Ναι, από ό,τι βλέπω το σημειώνω. Πριν δώσω το λόγο τώρα στους δύο εισηγητέ, ε, θα ήθελα να σας εξηγήσω λιγάκι μερικά πράγματα για το χρονοδιάγραμμα. Αυτό που διακυβεύεται για τις δύο αυτές υποθέσεις είναι το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης. Πρόκειται για έναν οριζόντιο μηχανισμό. Έχουμε τρία μέσα χρηματοδότησης που αναθεωρούνται. Είναι εκείνο της σταθερότητας, είναι το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι και το μέσο για τη συνεργασία με τις ε, βιομηχανημένες χώρες. Ξέρετε ότι υπάρχει ομάδα εργασίας όπου συμμετέχουν οι εισηγητές από τις τρεις επιτροπές που ασχολούνται με την εξωτερική δράση προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη θέση από πλευράς μας για το θέμα. Και μετά από πρόταση της ομάδας αυτής εργασίας, οι συντονιστές της δικές μας επιτροπής συμφώνησαν να έχουμε σύντομα μια δεύτερη ανάγνωση εδώ και μετά να υπάρξει ψηφοφορία το Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Γι' αυτό και η ψηφοφορία για αυτά τα θέματα στη δικιά μας Επιτροπή θα λάβει χώρα αύριο. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας και σε κάποιες διατάξεις πολύ αυστηρές που έχουν να κάνουν με το παραδεκτό των τροπολογιών σε δεύτερη ανάγνωση. Ο κανονισμός του Κοινοβουλίου, το άρθρο 66 παράγραφος 2, προβλέπει ότι οι τροπολογίες ε, του Συμβουλίου δεν είναι παραδεκτές παρά μόνο εφόσον συνάδουν με το άρθρο 156 και 157 και εφόσον επαναφέρουν τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ή καταλήγουν σε συμβιβασμό ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ή εφόσον τροποποιούν στοιχεία της πρότασης του Συμβουλίου, το οποίο όμως δεν υπήρχαν στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ή που είχαν διαφορετική φύση και που δεν τροποποιούν ουσιαστικά βάσει του άρθρου 159 ή αν πρόκειται αν πρόκειται για μια νέα θέση διαφορετική από εκείνη που είχαμε στην πρώτη ανάγνωση. Το ίδιο άρθρο λέει επίση ότι η απόφαση του Προέδρου για το παραδεκτό ή όχι των τροπολογιών ε, είναι οριστική η απόφαση αυτή. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη μετάφραση όμως. Επειδή πήγε το θέμα, δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί η μετάφραση της έκθεσης αυτής. Ε, ήταν έτοιμη σήμερα το πρωί μόνο. Τα δύο έγγραφα υπάρχουν σε 13 μόνο γλώσσες. Κύριε Μίτσελ, σας δίνω το λόγο παρακαλώ για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν ε, επιδιώκουμε τη μικροδιαχείριση, ούτε επικεντρωνόμαστε σε αποφάσεις επιμεμονωμένων προγραμμάτων και έργων οι τροποποιήσεις θα διασφαλίσουν ότι οι νομοθέτες θα διατηρήσουν τον έλεγχο επιστρατηγικών αποφάσεων. Τώρα, γιατί το θέλαμε αυτό. Το θέλαμε διότι θέλαμε να παίξουμε πιο αποφασιστικό ρόλο σε φύλακες, διασφαλίζοντας ότι οι βασικοί στόχοι θα χρηματοδοτούνται, όπως ορίζονται από τις συνθήκες αναπτυξιακή συνεργασία, μείωση και εξάλληψη της φτώχειας σε τελευταία ανάλυση. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό θέλουμε. Δεν είναι αυτά θέματα του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο φαίνεται ότι τώρα ε, συνεταιρίζονται κατά του Κοινοβουλίου και η Κομισιόν δεν ε, είναι δίκαιος παίκτης μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Πολλές φορές ε, ε, μιλούν με μια φωνή γιατί έχουν την Προεδρία. Και εμείς όμως μιλούμε με μια φωνή και η διάσκεψη των Προέδρων μας στηρίζει απόλυτα. Αγαπητή Πρόεδρε, το ταχύτερο περάσει αυτό από τη δεύτερη ανάγνωση και τη συνδιαλλαγή τόσο το καλύτερο, γιατί θέλουμε να διευκρινιστεί ότι όποια τροπή και να πάρουν τα πράγματα δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από τη θέση μας που έχει συνταγματική βάση και μας κάνει συνομοθέτες. Ευχαριστώ τα μέλη για την υποστήριξη, όχι μόνο εδώ, αλλά και σε όλες τις επιτροπές. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπουμε ότι μας υποστηρίζει η διάσκεψη των Πρόεδρων. Ας πάμε στη δεύτερη ανάγνωση και στην συνδιαλλαγή για να δούμε αν μπορεί να επιληθεί γρήγορα το θέμα. Ε, oui. Alors, monsieur, on m'informe que monsieur euh, a du ο κύριος Γκέρενς έχει καθυστερήσει από ό,τι μου λένε. Θα φτάσει στις 9-10 ε, παρατέταρτο. Φαίνεται ότι λόγω της κίνησης της Βρυξέλλες έχει μπλοκαριστεί και θα αργήσει. Συνεπώς, θα ξεκινήσουμε συζήτηση για την έκθεση Μίτσελ. Ο κύριος Μπέρμαν πρώτα έχει το λόγο. Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. η δημοκρατία ποτέ δεν θεωρείται δώρο. Πάντα ήταν αγώνας. Ο δημοκρατικός έλεγχος είναι κάτι που πρέπει κανείς να κερδίσει και να φροντίσει να το κρατήσει. Γι' αυτό και κάνουμε προσπάθειες. Πιστεύω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να μείνει σε αυτήν τη θέση με την οποία συμφωνεί και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει ο Γκί Μίτσελ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κέλλερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Μίτσελ και με τον κύριο Μπέρμαν και οι πράσινοι θα μείνουν σε αυτή τη θέση είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο έδωσαν τέτοια μάχη για τη συνθήκη της Λισαβόνας και πάντα το επιχείρημα ήταν ότι θα αυξάνονταν οι εξουσίες του Κοινοβουλίου και τώρα καταλήγουν ότι δεν θα μας δώσουν αυτή την εξουσία που είναι νόμιμο δικαίωμά μας, καλύπτεται από τη συνθήκη. Εκπροσωπούμε τους πολίτες και πρέπει να έχουμε λόγο σε θέματα στρατηγικής σημασίας και όχι να τα εξουσιοδοτούμε αναθέτοντας τα αλλού σε ανθρώπους που δεν έχουν έλεγχο, γιατί εμείς εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Καλό λοιπόν ε, να ακολουθήσουν όλοι την γραμμή πλεύσης του κυρίου Μίτσελ μέσα από αυτή τη σκοπιά. Ευχαριστούμε. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή, μήπως θέλουν να πάρουν το λόγο για τη δεύτερη αυτή ανάγνωση. Παρακαλώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σημειώσαμε την θέση της Επιτροπής σας για τη δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης Μίτσελ και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει για την έκθεση Γκούρενς, μια που οι τροπολογίες έχουν να κάνουν με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της δεν μπορεί παρά να επαναλάβει τη θέση της, έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. Δηλαδή, οι τροποποίησεις των κανονισμών που έχει υποβάλει η Επιτροπή είναι τροποποίησης κανονισμού μέσω συνεργασίας για ε, ανάπτυξη του 2006. Πρόκειται για κανονισμό ήδη πάρα πολύ πυκνό που προέβλεπε ήδη πολλούς προσανατολισμούς στρατηγικής σημασίας όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων. Και πολύ συγκεκριμένα έλεγε τα κονδύλια αυτά με ποιο τρόπο μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Συνεπώς, στο στάδιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι όπως έχει σήμερα ο κανονισμός DCI, δεν μπορεί παρά να επαναλάβει τη θέση της. Υποστηρίζει δηλαδή ότι τα έγγραφα για τη στρατηγική αναχώρα και τα πολιετή σχέδια στα πλαίσια τα θεματικά δεν μπορούν να θεωρηθούν κατ' εξουσιοδότηση πράξη, νομοθετικές πράξεις δηλαδή, αλλά εφαρμοστικές. Και αυτό οφείλεται, όπως έλεγα και πριν, στο γεγονός ότι το μέσο συνεργασίας για ανάπτυξη είναι ένας πολύ πυκνός κανονισμός με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Από τη δικιά μας την πλευρά αυτό που θέλουμε πάντως να καταδείξουμε είναι ότι υπάρχει κάτι που επήγει και πήγη για τις χώρες παραγωγούς μπανάνας που βρίσκονται σε μια αρκετά δύσκολη θέση σήμερα και που θα θέλανε τα κονδύλια αυτά ήδη από πέρυσι να είχαν απελευθερωθεί. Για τις χώρες ΑΚΕ λοιπόν από πλευρά της Κομισιόν γίνονται διαβήματα. Δεν ξέρω αν το ίδιο γίνεται και από το Κοινοβούλιο. Σας το λέω πάντως για να σας δείξω πόσο πολύ επίγει η κατάσταση για τις χώρες ΑΚΕ που κατά κάποιο τρόπο είναι όμοιροι τώρα αυτής της κατάστασης. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το ότι όταν είχαμε την πρώτη ανάγνωση εμείς κάναμε μια μεταβατική πρόταση η οποία θα έπρεπε να καλύπτει την περίοδο από σήμερα, από την έγκριση δηλαδή αυτών των δύο κανονισμών και το νέο πολιετές ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ήτανε ε, μόντως βιβέντη λύση, η οποία όμως θα διασφάλιζε αυτό που ζητάει τώρα το Κοινοβούλιο, δηλαδή την εφαρμογή, την καλύτερη εφαρμογή με περισσότερες λεπτομέρειες και σε βάθος του ορισμού των στρατηγικών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει την πρόταση αυτή ακριβώς για να προσπαθήσει να καλύψει τα τρία αυτά χρόνια σχετικά με το DCI. Και πρότεινε και γενικές αρχές που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ε, με το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο που βέβαια βρίσκεται σήμερα σε πολύ αρχικό στάδιο για να μπορούμε από τώρα να πούμε ποια θα είναι τα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο κατά εξουσιοδότηση πράξεων. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλετε, έδειξε την καλή της θέληση, έδειξε τη θέλησή της για συμβιβασμό. Από εδώ και πέρα, στο ίδιο πνεύμα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε προκειμένου να εξευρεθεί γρήγορα μια λύση. Μια λύση μάλιστα που δεν θα ζημιώσει τους εταίρους μας από τις χώρες ΑΚΕ, που έδειξαν την εμπιστοσύνη τους εμάς στις διαπραγματεύσει της Γενέβης και που τώρα αναγκάζονται να πληρώσουν μια τιμή που τους επιβάλλεται για λόγους που στο κάτω-κάτω δεν τους αφορούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κύριε Μίτσελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τη θέση της αυτή. Σημείωσα τις ε, λέξεις ταχεία απόφαση και η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι χώρες ΑΚΕ. ως ε, ομάδα χωρών ε, που θα προβληθούν ιδιαίτερα για ε, στα πλαίσια του ρόλου μας ως συνομοθέτη. Θα ήθελα να πω, και το έχω ξαναπεί, εγώ στη χώρα μου, ε, όταν εξηγούσα στην προεκλογική εκστρατεία της συνθήκη της Λισαβόνας, τους έλεγα ότι θα ενισχυθεί η διαφάνεια ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην κοινή λήψη αποφάσεων. Αυτό εξασφαλίζει η συνθήκη, αυτό ζητάμε. Και υπάρχει πρόβλημα ε, όταν δεν δείχνουν τα δύο άλλα θεσμικά όργανα σεβασμό στο Σύνομο Θέτη. Όταν με απαντήσεις θα πρέπει να εξετάζονται από τα άλλα θεσμικά όργανα βάσει της συνθήκης. Πάμε λοιπόν, ας πάμε στη δεύτερη ανάγνωση το ταχύτερο δυνατόν και στη συνδιαλλαγή, να δούμε αν μπορεί να λυθεί το θέμα, να ξέρουν όλοι που βρίσκονται. Και θα ήθελα να πω στην Κομισιόν, παρακαλώ, αρχίσετε να παίζετε το συνταγματικό σας ρόλο ως το θεσμικό όργανο που σκοπό έχει να συμβάλλει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο αρμοδίων για την νομοθεσία οργάνων. Ε, γιατί αλλιώς πραγματικά χάνονται ε, σκληρές προσπάθειες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκέρενς δεν φτάσει ακόμη. Θα έλεγα να διακόψουμε την εξέταση αυτού του σημείου και να περάσουμε στο επόμενο που προβλέπει η μερίσια διάταξη. Θα έχουμε παρουσίαση από την συνάδελφο, την κυρία Τσίμερ, της έκθεσής της. Έκθεση που αφορά την επισητιστική ασφάλεια και το νέο στρατηγικό πλαίσιο που προτείνει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Τσίμερ που ή άλλως είναι συγκήτρια για αυτή την έκθεση και η οποία έχει προσκαλέσει εκπρόσωπο του δικτύου Άπροντερ που και εκείνο θα μας κάνει κάποια σχόλια μια παρουσίαση. Κυρία Τσίμερ, να μας παρουσιάσετε πρώτα το έγγραφο εργασίας σας που θα χρησιμοποιηθεί ως ε, υλικό για την έκθεση αυτή καθ' αυτή. Έχετε 10 λεπτά κυρία Τσίμερ. Yeah, vielen Dank, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση που θέλω να θέσω προσυζήτηση με έγγραφο εργασίας στην Επιτροπή μας στηρίζεται σε δύο ανακοινώσεις της Κομισιόν από τον περασμένο Μάρτιο που έχουν στενή σχέση μεταξύ τους αλλά συνειδητά δεν έχουν συνδεθεί η μία με την άλλη για να είναι σαφές ότι και οι δύο εκθέσεις, οι δύο ανακοινώσεις μάλλον της Κομισιόν ε, έχουν παρόλα αυτά διαφορετικό προσανατολισμό. Πρόκειται αφενός για την ανακοίνωση της Κομισιόν για το πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, υποστήριξη των αναπτυσσομένων χωρών ώστε να βελτιώσουν την επισητιστική ασφάλεια και το δεύτερο, η δεύτερη ανακοίνωση της Κομισιόν αφορά κυρίως την ανθρωπιστική βοήθεια στον επισητιστικό τομέα. Με βάση το έγγραφο εργασίας που έδωσα προς συζήτηση εδώ και που αποτελεί και βάση για το προσανατολισμό μου κατά την επεξεργασία της έκθεσης, θα ήθελα να τονίσω τα εξής. Πρώτον, πιστεύω ότι ιδιαίτερα η ανακοίνωση της Κομισιόν για την βελτίωση της επισητιστικής ασφάλειας πολύ σωστά στηρίζεται σε τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένους πυλώνες και μέσα σε αυτά τα πολιτικά πλαίσια επιχειρεί να υποβάλει προτάσεις για τις οποίες νομίζω ότι βελτιώνουν ε, την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια. Όμως, από αυτές τις πληροφορίες λείπει μια ευρύτερη προσέγγιση για την εξέταση της επισυδιστικής κρίσης, ιδιαίτερα το 2008. Καταρχήν, θα πρέπει να δούμε το γενικότερο θέμα της αντιμετώπισης του θέματος βελτίωσης της επισητιστικής ασφάλειας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επιχειρήσουμε και αναφέρεται βέβαια κάπως, αλλά θα πρέπει να Κρίνομαι γιατί και να αποφασίσουμε γιατί το 2008 προέκυψε η κρίση στην επισητιστική ασφάλεια. Αυτό λείπει. Έχουμε παραγνωρίσει κάτι που είναι κεντρική σημασίας και έτσι η ανακοίνωση της Κομισιόν ε, καταλήγει να είναι πολύ στενή στην προσέγγιση της. Αυτό θα το επιχειρηματολογήσω. Καταρχήν ε, συμφωνούμε διότι στην ανακοίνωση της Κομισιόν γενικά γίνεται μια αναφορά στην, στον ασταθή εφοδιασμό τροφίμων που αποτελεί μια πρόκληση για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια περιοχή της ε, Αφρικής και τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η ΦΑΟ όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ανακοινώνει ότι το 2010 ε, οι άνθρωποι που πεινούν ανέρχονται σε 925 εκατομμύρια και υπάρχουν πολύ περισσότεροι υποσυτιζόμενοι τώρα από ότι, για παράδειγμα, στην αρχή της τωρινής κρίσης. Αυτό που λείπει όταν πρόκειται για την περιγραφή του προβλήματος αλλά και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων μας είναι πρώτον μια εκτίμηση ότι η οξία κρίση, η παγκόσμια επισητιστική κρίση του 2008 οφείλεται σε αποθέματα περιορισμένα, σε κρίση στη συγκομιδή, τότε δεν ε, υπήρχαν αρκετά αποθέματα. Αυτό όμως δεν είναι ο μόνος λόγος, αφού δεν αναφέρεται ιδιαίτερα η ε, παραγωγή τροφίμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΠΑ και βέβαια το πρόβλημα των βασικών τροφίμων αλλά και πρώτων υλών. Ε, εδώ παραπέμπω και στη φούσκα των πρώτων υλών. Σε σχέση με την, και σε συνδυασμό με την ε, αύξηση του πληθυσμού, το αποτέλεσμα ήταν ότι πάλι ε, τέθηκε ένα αμφιβόλο η επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Κομισιόν στην προσέγγιση της αναφέρεται στο γενικότερο θέμα της έλλειψης ασφάλειας στον επισητιστικό τομέα και θίγει και διεθνή θέματα όπως αυτά ανέκυψαν, αλλά ε, δεν ε, αναλύει επαρκώς την κρίση του 2008 και τα αίτια της και δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε, ώστε τέτοιες οξύες κρίσεις να μην επαναληφθούν. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω αυτή την αμφισημία. Επίσης επισημαίνω ότι παρά των τωρινών υποθέσεων των οικονομολόγων σχετικά με το θέμα της μεγάλης διακύμανσης των τιμών των τροφίμων, οι τεράστιες αυξήσεις των τιμών δεν οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής στις χώρες του Νότου, αλλά σε αύξηση της γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη και της ΗΠΑ. Και εδώ είναι η σημαντικότερη κριτική που θέλω να εκφράσω και που θα τη συνεχίσω κατά τη συζήτηση με τους συναδέλφους και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους ειδικού τις επόμενες εβδομάδες και τους μήνες. Χρειαζόμαστε σαφέστερη περιγραφή του τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξαντλήσει τα περιθώρια που έχει. Θεωρώ ότι οι προτάσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν ε, θα πρέπει να είναι επαρκής, ούτως ώστε να παρεμποδίζουν τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Τέτοιες εξελίξεις δηλαδή, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, θα πρέπει να επηρεάζονται μέσα από τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι θεωρώ πως λείπει μια ε, συγκεκριμένη σύνδεση, τουλάχιστον στην πρώτη ανακοίνωση, που αναφέρεται στο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των αναπτυσσομένων για τη βελτίωση της επισητιστικής ασφάλειας, διότι εκεί δεν φωτίζεται παρκώς η σχέση που υπάρχει μεταξύ κλιματικής αλλαγής, των, της ε, ανάγκης και έλλειψης τροφίμων και των μεταναστευτικών ροών, ροών και εσωτερικής μετανάστευσης αλλά και μετανάστευσης από ε, τη μία Ήπειρο στην άλλη. Στην άλλη ανακοίνωση, η οποία αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια στον επισητιστικό τομέα, εκεί καλύτερα αναφέρονται τα συγκεκριμένα μέτρα, χωρίς να αναπτύσσονται πολύ, αλλά πάντως ε, είναι σαφή, ε, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η πρώτη ματιά στα απαραίτητα μέτρα. Είναι λοιπόν απόλυτα θεμητό το γεγονός ότι επέλεξαν να υποβάλουν δύο διαφορετικές ε, ανακοινώσεις. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι, ποιο είναι το σημείο κινήσεως, ποιο είναι το πρίσμα μέσα από, τα οποία, μέσα από το οποίο βλέπουμε τα πράγματα και ποιος είναι ο προσανατολισμός μας για την ανάληψη δράσης. Τώρα, το έγγραφο εργασίας περιέχει σειρά θέσεων που ως επιτοπλίστων ε, αναφέρονται στους τέσσερις πυλώνες. Στην πρώτη ανακοίνωση η Κομισιόν συμφώνησε και σχολιάζει τα μέτρα αυτά. Συμφωνούμε και θεωρούμε όμως ότι υπάρχουν ανάγκες για διευκρινήσεις και προσθήκες. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη νέα ημερήσια διάταξη για την επισητιστική ασφάλεια. Εγώ χαίρομαι διότι η Κομισιόν θεωρεί ότι χρειάζονται στη γεωργία και την επισητιστική ασφάλεια μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ε, οι δαπάνες από το 17% στη Γεωργία το 80% έπεσαν στο 5% και αυτό συνιστά μείζον πρόβλημα και βέβαια προγράμματα βοήθειας περιφερειακά, εθνικά για την υποστήριξη της Γεωργίας είναι απαραίτητα ώστε και να εντάξουμε εδώ και τη γενικότερη στρατηγική καταπολέμηση της φτώχειας. Για τη διαθεσιμότητα των τροφίμων πολύ σωστά αναφέρεται ότι ο ΦΑΟ περιμένει η ανάγκη για γεωργικά προϊόντα ε, να θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2017. Αυτό δεν αναφέρεται μόνο στην αύξηση τη δημογραφική, αλλά και την ποιότητα και την ε, σύνθεση των τροφίμων, δηλαδή την θρεπτική τους αξία και τις σχετικές ε, προσδοκίες. Οι προσεγγίσεις μας εδώ θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές και οικολογικά διατηρήσιμες, βιώσιμες και να ε, στηρίζονται σε χαμηλό εξωτερικό input. Θα πρέπει να έχουμε γι' αυτό πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες, την πρόσβαση στην αγορά, έρευνα και ε, υποστήριξη των μικρών γεωργών. Σε αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό ότι η Κομισιόν σαφώς επισημαίνει ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει μαζικά να υποστηριχθούν, γιατί μεταξύ άλλων αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής της Κομισιόν, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, ιδιαίτερα στο μέλλον. Θα ισχύει αυτό, δηλαδή, ακόμη περισσότερο. Επίσης, λείπει το γεγονός ότι στα πλαίσια της συζήτησης και στα πλαίσια της πρότασης της Κομισιόν ε, λείπει λοιπόν μία αναφορά στις επίκαιρες συζητήσεις που γίνονται τώρα και που ξεπερνούν το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας, food security. Θα ήθελα να τεθεί τουλάχιστον και ένα ακόμα θέμα, όπως π.χ. σε ποιο βαθμό είναι σωστό να συζητήσουμε και το θέμα της επισητιστικής κυριαρχίας. Δηλαδή να δούμε και σε επίπεδο περιφερειακό αλλά και γενικότερο το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας πέρα από εθνικά σύνορα. Ίσως θα έπρεπε και αυτό να συμπεριληφθεί στη συζήτηση που κάνουμε εδώ όλοι μαζί. Και αυτή η προβληματική πρέπει να ανοίξει και σε σχέση και εν ώψη της ακρόασης που θα οργανώσει τον Ιούνιο νομίζω εδώ το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, προς το παρόν αφήνω κατά μέρος τα άλλα θέματα που αναφέρονται στους τέσσερις πυλώνες για να τονίσω κάποια επιμέρους προβλήματα που πιστεύω ότι πρέπει σε αυτά να εστιάσουμε περισσότερο. Πρώτον, το θέμα της διακύμανσης των τιμών των τροφίμων και της κερδοσκοπίας που γίνεται στα τρόφιμα. Το Δεκέμβριο του 2010, ο δείκτης τιμών τροφίμων ήταν στα 215, ένα, κατά ένα μόριο χαμηλότερο από το υψηλότερο σημείο στο οποίο έφτασε κατά την επισητιστική κρίση. Η κερδοσκοπία παίζει μεγάλο ρόλο και επηρεάζει τις τιμές. Αυτό έγινε και το 2008 αλλά και τώρα ε, που αυξήθηκαν πάλι οι τιμές των τροφίμων. Ένα άλλο πρόβλημα που θέλω επίσης να αναφέρω είναι το ε, θέμα του land scrubbing. Καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας ότι 33 εκατομμύρια εκτάρια γη απο, αγοράστηκαν από ξένους επενδυτές και έτσι δεν προωθείται ο εφοδιασμός στις χώρες αυτές. Εκεί δηλαδή στις χώρες όπου το επισητιστικό πρόβλημα είναι ε, μεγάλο στη Σαουδική Αραβία 1500, στην ε, Τανζανία, στη Σαουδική Αραβία, στο Σουδάν αγοράστηκαν ε, εκατοντάδες στρέμματα. Ε, αυτό δημιουργεί πρόβλημα και για τις μικρές ε, αγροτικές οικογένειες, αλλά δημιουργείται και πρόβλημα μεταξύ χωρών, γιατί έτσι γίνεται μετεγκατάσταση και ε, μετακίνηση των αγροτών που χάνουν την ε, γη τους και τη δυνατότητα παραγωγής. Σταματώ λοιπόν στο σημείο αυτό. για την ανακοίνωση της Κομισιόν για την ανθρωπιστική βοήθεια. Τονίζω ότι είναι σημαντικό η σύμβαση, να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση για την επισητιστική βοήθεια ε, βασίζεται στη δεκαετία του 60 και δεν ανταποκρίνεται πια στις ε, απαιτήσει ε, όπως διαμορφώθηκαν για τον επισητιστικό εφοδιασμό και νομίζω ότι οι νέες αυτές διαπραγματεύσεις είναι πολύ σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και εδώ να παίξει το ρόλο που της αρμόζει. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμός με άλλους φορείς για την επισητιστική ασφάλεια, χρειάζεται καλύτερο συντονισμός των χρηματοδοτικών μέσων, η διακυβέρνηση επίσης θα πρέπει και η σύμβαση, όπως είπα, θα πρέπει να επανεξεταστεί και χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια της λήψης αποφάσεων για καλύτερο monitoring, έλεγχο, παρακολούθηση και σίγουρα, σίγουρα θα πρέπει να επιβάλλουμε και συγκεκριμένες ε, διασφαλίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σημαντικότατο έργο και που για τη δική μας την Επιτροπή ως ζήτημα βρίσκεται μεταξύ των πρώτων μεριμνών μας. Και τώρα η κυρία Ιλμερ από την Άπροντεφ για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σχολιάσω την έκθεση και το θέμα αυτό, την έκθεση της κυρίας Τσίμερ. Είμαστε μέλη των ε, βασικών περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Ευρώπη και θέλουμε να αναπτύξουμε τρία βασικά σημεία. Γιατί η ανακοίνωση για την επισητιστική ασφάλεια και τη σχετική στρατηγική και πρόγραμμα είναι μια έμεση απόκριση στην ε, κρίση των, της αγοράς των τροφίμων. Εδώ καλωσορίζουμε τη βασική σύσταση να επικεντρωθούμε και να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στους μικρούς γεωργούς ως μέρος της λύσης για την επισητιστική κρίση. Καλώς υπάρχει μνήμα στην οικολογική αποτελεσματικότητα και την διαφοροποιημένη λειτουργία της γεωργίας. Εδώ οι κοινωνικές λειτουργίες και η κοινοτική προσέγγιση στην παραγωγή τροφίμων είναι σημαντική. Ως προς την στρατηγική επισητιστική ασφάλεια, ε, εδώ το τι είδου τεχνολογικά μέσα και τι είδους πρακτικές θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη είναι ένα ζήτημα. Και εδώ θα πρέπει να συνδυάσουμε την έρευνα για την ε, γεωργία με τις επιπλέον γνώσεις που διαθέτουμε. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε να μην υποστηρίξουμε τεχνολογικά μέσα που δεν είναι βιώσιμα. Επίσης, ε, τα πορίσματα της έρευνας Άιστατ είναι πολύ σημαντικά για τον συνδυασμό γνώσης έρευνας ε, και έρευνας στην γεωργία έχουμε δώσει έμφαση στο ότι η βιοπικιλότητα και η φυσική πόρη, καθώς και το να την υπόψη τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά για να ενισχυθεί η παραγωγή των μικρών γεωργών. Για τα εξωτερικευμένα μοντέλα αγροτική παραγωγής, εδώ θέλουμε να αποφύγουμε τα συνθετικά λοιπάσματα και ζυζανιοκτώνα ε, ως εξωτερικά ε, στοιχεία της ε, γεωργίας και ως αρνητικά αποτελέσματα να προάγουμε την χρηστή διαχείριση των υδάτων και την μεθοδική χρήση των λιπασμάτων. Τα στοιχεία Αυτά συνδυάζονται με, με σωστές πρακτικές ε, της αγοράς και σωστές εμπορικές συμπεριφορές, προκειμένου να έχουμε παραγωγικότητα και εισόδημα. Αυτό το στηρίζουν πολλές μελέτες με κυβερνητικό οργανώσεων σε πολλές χώρες και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως ε, το Πανεπιστημίο του Cambridge και της αρμόδιας ε, μονάδας του, και Επίσης όλα αυτά θα συνεισφέρουν και ως ανταπόκριση στις κλιματικές αλλαγές, τον μετριασμό των φαινομένων, την χαμηλότερη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, την ανθεκτικότητα των, ε, ε, των ε, καλλιεργιών, την λειψιδρία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Συστήνουμε λοιπόν και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της επιστημιστικής κρίσης. Η πράσινη επανάσταση είναι κάτι που θέλουμε να ενθαρρυνθεί. Έχουμε δει το παράδειγμα της Ασίας που είναι αρνητικός προς τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική προστασία και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα καθώς και το εισόδημα των γεωργών. Τώρα μερικά σχόλια για την έκθεση της κυρίας Τσίμερ. Καλωσορίζουμε την ανακεφαλαίωση των χαμένων ευκαιριών που οδήγησαν στην επιστημιστική κρίση. Υπάρχουν και αθέμετοι όροι ανταγωνισμού. Είναι και αυτός ένας λόγος που προέκυψε η κρίση αυτή. Θα πρέπει να αυξήσουμε την επιστημιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες θα πρέπει να διευκολυνθούν να καταρτήσουν δικέ τους στρατηγικές. Για την αγορά και την διακύμανση, την έντονη διακύμανση των τιμών, αυτό έχει να κάνει και με την κερδοσκοπία στα βασικά αγαθά, όπως επισημαίνει και η έκθεση Θήμερ, και τα χρέη που υπάρχουν στον γεωργικό τομέα. Οι πιο ευάλωτες ε, χώρες είναι αναπτυσσόμενες και ιδίως στον αγορά των τροφίμων τους θα πρέπει να μπορούν να προστατεύσουν τα δικά του συστήματα παραγωγή τροφίμων και τι δικέ του αγορέ. Δεν θα πρέπει να του ασκούνται πιέσει να ε, επαφίενται σε αγορές ασταθείς για τη δική τους προμήθεια σε τρόφιμα, αλλά να έχουν ένα αποτελεσματικό δικό τους σύστημα. Για τα αναποτελεσματικά μέτρα, και αυτόν η ευθύνη αναφέρεται στην έκθεση Τσίμερ, Υπάρχουν πολλές επιλογές και ευκαιρίες στο να έχουμε μία προσέγγιση πιο στοχευμένη, ε, με λιγότερα εξωτερικά αποτελέσματα και να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα των ε, φύλων ε, με το σύστημα τοπικών κοινοτήτων, με την παροχή υπηρεσιών, την ενίσχυση των οργανώσεων γεωργών και με ερευνητικά προγράμματα που να παρακολουθούν τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και ιδίως τις παραδοσιακές γνώσεις αναφύλλω και την τεχνογνωσία για την βιοπικιλότητα, για την αρπαγή ε, εδαφών και τις διαφορές ε, περί γεών, εδώ τα βιοκαύσιμα και η αρπαγή γεών ε, έχει οδηγήσει σε ανταγωνισμό για τα γεωργικά εδάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τον αναδασμό ή τουλάχιστον επιτρέψει τον αναδασμό σε αναπτυσσόμενε χώρε όπου έχουν αναλυθεί τέτοιε πρωτοβουλίε. Πιστεύουμε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ότι θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση του και στι αναπτυσσόμενε χώρε, γιατί έτσι παρουσιάζονται και οικονομικέ ευκαιρίε και θα πρέπει να υποφεληθούν οι χώρε αυτέ. Για τι ευρωπαϊκέ ε, πρακτικέ κατανάλωση ε, θα πρέπει. να συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσίμερ, ευχαριστώ για το σχέδιο αυτό. Ε, έχει, προχωράει πολύ σε ορισμένα σημεία, αλλά γενικά είναι καλό. Ευχαριστώ πολύ και για τη συμπερίληψη της συνοχής στην πολιτική μας. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, για τις επιδοτήσεις στο γεωργικό τομέα. Και εγώ με πολύ κριτικό μάτι τις αντιμετωπίζω αυτές τις επιδοτήσεις, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές μας εν ώψη της σημερινής κατάστασης της Αφρικανικής Γεωργίας ιδιαίτερα ε, και στην Ασία, θα, θα βοηθούσε ιδιαίτερα και την Ασία και τη Λατινική Αμερική και νομίζω ότι αυτή την πρόκληση θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μαζί με τις αφρικανικές χώρες. Δεύτερον, για την κριτική της εμπορικής στρατηγικής που τη θεωρώ θεμητή κριτική. Νομίζω ότι η αηφορία, η βιωσιμότητα επικεντρώνεται πολύ στην περιβαλλοντική πολιτική παραγνωρίζοντας πτυχές κοινωνικές και οικονομικές. Είναι σημαντικό οι αναπτυσσόμενοι, οι εταίροι μας, να έχουν περιθώριο ελιγμών μεγαλύτερο για να διασφαλίζουν την επισητιστική ασφάλεια και κατά δεύτερο λόγο, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να τονιστεί περισσότερο, ε, για να δημιουργούν τοπικές και περιφερειακές αγορές για να προάγεται το εμπόριο μεταξύ νοτίων χωρών. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέση έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ να χαιρετήσω την ε, κυρία Σίμερ για το έργο τη και πολύ σύντομα να πω ότι στηρίζω τι κεντρικέ ιδέε τη εκθεσή τη. Δηλαδή ότι ο ρόλο μα ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ε, κατά το μέγιστο βαθμό να εξασφαλίσουμε την επιβίωση και την ε, λειτουργία των μικρών παραγωγών. Επίση την πρόσβαση στα εδάφη του, την δυνατότητα να αναπτυχθούν, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Ε, νομίζω ότι εκεί υπάρχει έλλειμμα στην ανάπτυξη και στην επισητιστική ασφάλεια και την ε, κυριαρχία. Αυτές, ε, αυτά τα δύο στοιχεία είναι οι απαντήσεις στο πρόβλημά μας. Η τοπική παραγωγή και όχι μόνο η γεωργία για σκοπούς εξαγωγών. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ενδογενής ανάπτυξη Δηλαδή, να εφαρμόσουμε μια τέτοια έννοια όχι μόνο στην Αφρική και την Ασία αλλά και στην Ευρώπη. Και επιπλέον μια ιδέα που θέλω να στηρίξω μέσα από αυτή την έκθεση αυτή είναι ότι και για μας αποτελεί αυτό μέρημνα ε, η αρπαγή γεών από τρίτε χώρε είναι κάτι που ανησυχεί. Όπω ε, η Νότια Κορέα. Ένα παράδειγμα πολύ αρνητικό και θα πρέπει να μας απασχολήσουν και τέτοια ζητήματα πολύ ανησυχητικά για, την ε, μελλοντική, ε, για τις μελλοντικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ο κύριος Νόισερ. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια, την κυρία Τσίμερ για την ε, εκτενή και λεπτομερή της έκθεση. Εγώ θα κάνω μια διευκρίνηση που αφορά την κερδοσκοπία στα τρόφιμα. Στο Βερολίνο έχουμε τώρα τη λεγόμενη πράσινη εβδομάδα. 48 Υπουργοί Γεωργίας συμμετέσχουν. Αυτοί οι 48 Υπουργοί Γεωργίας βλέπουν παρόμοιο κίνδυνο ε, σήμερα όπως και το 2008 με έκρηξη των τιμών των γεωργικών προϊόντων και κερδοσκοπία στις πρώτες ύλε. Οι 48 Υπουργοί Γεωργίας κάλεσαν τους G20 και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο πρέπει να κάνει. Κάλεσαν λοιπόν τους G20 να φροντίσουν για μεγαλύτερη διαφάνεια ε, στα χρηματιστήρια. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι κερδοσκόποι στα γεωργικά προϊόντα είναι γεωργοί, είναι ε, χρηματιστηριακοί κύκλοι, είναι η παραγωγή ε, των τροφίμων, των επεξεργασμένων προϊόντων. Χρειάζεται ασφάλεια. Η εξεγέρσεις στην Αλγερία και την Τινησία πρόσφατα αφορούν επίσης και τις αυξημένε τιμές στα τρόφιμα, τα γεωργικά προϊόντα και βλέπουμε με, με τα παραδείγματα αυτά πόσο ευαίσθητο θέμα είναι αυτό των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Ο Πασκάλ Λαμίου, Γενικός ε, Διευθυντής του ΠΟΕ, λέει ότι στα σιτηρά και τον αραβόσιτο ε, οι τιμές ε, έφτασαν και ξεπέρασαν σε ορισμένες χώρες ε, τις τιμές του 2008. Μετά από αυτό πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή ενός παγκοσμίου συστήματος αποθεμάτων για τα βασικά γεωργικά τρόφιμα τουλάχιστον. Ευχαριστούμε κύριο Κάσμαρεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να προσθέσω τι δικέ μου ευχαριστίε, τι ευχαριστίε των υπολείπων για την κυρία Τσίμερ. Είναι σημαντικό ε, το θέμα αυτό και ιδίω μια πτυχή του που συζητιέται και στο έγγραφο. Ιδίω λοιπόν το θέμα τη μελλοντική μεταρρύθμιση τη ε, κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή τη στιγμή οργανώνονται πολλέ διαβουλεύσεις, ε, διασκέψει, συζητήσει σε επίπεδο Γενική Διευθύνση Άγκρη. η σφαιρική προσέγγιση του θέματος της γεωργικής παραγωγής, αυτό το ζήτημα δεν συζητιέται επαρκώς. Με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος, δεν υπάρχει μετάφραση προς τα αγγλικά. Για κάποιο λόγο δεν ακούστηκε σωστά η αγγλική διερμηνία από ό,τι φαίνεται. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα γίνεται Συνεχώ συζήτηση για το μέλλον τη κοινή αγροτικής πολιτική. Και στο επίπεδο τη δική μα τη επιτροπή. Όμω δεν συζητάμε ακόμη για μια σφαιρική προσέγγιση τουλάχιστον όσο χρειάζεται για την κοινή αγροτική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που και σήμερα αναφέρθηκαν. Είναι δική μας η ευθύνη και αρμοδιότητα, διότι αν όλα αυτά παραμεληθούν, και αγνοηθούν, δεν θα καταλήξουμε σε σφαιρική προσέγγιση. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Κέλλερ για τη σφαιρική προσέγγιση στη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ μην ξεχνάμε τι είπε ο Επίτροπο για τη μεταρρύθμιση αυτή και την αναπτυξιακή τη διάσταση. Είπε και παραθέτω εδώ ότι πέρα από τι επιδοτήσει για τι εξαγωγέ, η ΚΑΠ δεν θα έχει καθόλου εξωτερικέ διαστάσει. Άρα, η εξωτερική διάσταση τη ΚΑΠ ε, θα έχει μηδενικό αντίκτυπο, όπω είπε και ο ίδιο. Πέραν από τι εξαγωγικέ επιδοτήσει δεν θα έχει κανένα. Καμία τέτοια διάσταση. Άρα, δεν μα μένουν και πολλά να κάνουν. Και για την αναπτυξιακή προοπτική το αν συμφωνεί μαζί μα ο Επίτροπο ή όχι είναι ένα θέμα. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι πτυχέ αυτέ και τα αποτελέσματα τα ενδεχόμενα τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ από αυτή την προοπτική. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η Επιτροπή ο κύριος Βιν... Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε και για αυτή την έκθεση που είναι εξαιρετική αντίδραση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανακοινώσεις θα έπρεπε να πω, γιατί είναι δύο ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν εδώ και ένα χρόνο. Η μία για την επισητιστική ασφάλεια και η άλλη για την ανθρωπιστική βοήθεια από τους συναδέλφους ε, της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης. Η κοινή δημοσίευση αυτή σκοπό είχε να έχουμε καλύτερη συνεργασία στην διαπαθή για την αντιμετώπιση της κρίσης και την επιστημιστική ασφάλεια και τις σχετικές τους πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μία από τις πτυχές που προσπαθήσαμε να καλύψουμε. Καθώς και οι διάφορες προκλήσεις, ο κατεπήγων χαρακτήρας και οι αποκρίσεις που χρειάζονται στις αναπτυξιακές μας επαφές. Να αντιδράσω κατά πρώτον σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση για την επισητιστική ασφάλεια αρχικά προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στην κρίση του 2008 με τρόπο σφαιρικό και να φέρουμε πάλι το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας στην προσοχή του κοινού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να ετοιμάσει την ανακοίνωση αυτή για διαφορετικούς λόγους. Και Κυρίως ήθελε να ενισχύσει τις γνώσεις μας, ώστε να ξέρουμε πώς να ε, αντιδράσουμε σε τέτοια ζητήματα επισητιστικής ασφάλειας και ιδίως ε, στα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών. Μια από τις πηγές εμπνευσής μας ήταν και το έργο της ε, IAS, ID. E e ε, της πολύ πυκνής ε, αυτής έκθεσης, ε, της μεστής ενόημα έκθεσης, για τα θέματα της επιστημιστικής ασφάλειας. Το θέμα της, των τροφίμων, των θρεπτικών στοιχείων των τροφίμων, των βιοκαυσίμων, είναι στοιχεία που καλύπτονται από την έκθεση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάσαμε την ανακοίνωση αυτή και όχι μόνο για τη διάσταση που αφορούσε την κρίση αυτή καθ' αυτή. Πολλοί ανέφεραν ότι υπάρχουν ε, ελλείψεις στην ε, ανακοίνωση, ίσως δεν είναι αρκετά επίκαιρη, βέβαια έχει περάσει και ένας χρόνος. Όμως να μην ξεχνάμε ότι η ανακοίνωση αυτή συνοδεύτηκε από ένα έγγραφο εργασία. Ε, πιο λεπτομερές, όπως το δικαίωμα των καταναλωτών στη, στα θρεπτικά στοιχεία, το θέμα της έντονης διακύμανσης του τιμών, τα θέματα πρόσβασης στη γη, Ακούσαμε επίσης κάποιες παρατηρήσεις για την επισητιστική κυριαρχία. Όπως έχω πει και σε άλλες ευκαιρίες, ως τώρα έχουμε προτιμήσει τον όρο επισητιστική ασφάλεια. Θεωρούμε ότι είναι πιο ε, κατάλληλος όρος και διεθνώς αποδεκτός Ω προ το νόημά του, ενώ η κυριαρχία είναι μια έννοια που σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Πιο δύσκολο να αντιληφθεί κανεί τι εννοούμε. Παρόλα αυτά, πολλές από τις πτυχές που καλύπτει ο όρος επισητιστική κυριαρχία ανακύπτουν και στην ανακοίνωση, αν και δεν χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό καθεαυτό ούτε τι ίδιε διατυπώσει. Πολλέ παρατηρήσει έγιναν για την έντονη διακύμανση των τιμών και τα αίτια αυτού του φαινομένου. Πράγματι, δεν έχουν αναλυθεί επαρκώ όλα τα αίτια στο έγγραφο εργασία που σα υπέδειξα. Προσπαθήσαμε να ανακεφαλαιώσουμε κάποιου παράγοντε ε, μια-δυο σελίδε, όμω, εάν δούμε τι συνέβη το 2008, και το τι συμβαίνει σήμερα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε κυρίως να αντλήσουμε διδάγματα. Ένα από αυτά είναι ε, μια συστηματική, ένα συστηματικό συνδυασμό πολλών διαφορετικών παραγόντων. Ένα, η αύξηση των τιμών και δεύτερο, η έντονη διακύμανση. Η κερδοσκοπία φαίνεται επίσης να είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Ένα από του παράγοντε για του οποίου γίνονται ακόμη έρευνε και μελέτε. Αυτή τη στιγμή, χωρί σαφή εμπεριστατωμένα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να αποφανθούμε ότι, ότι αυτό είναι το πρωταρχικό αίτιο, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ε, ο ρόλος της κερδοσκοπίας είναι καθοριστικός. Και το αντίστροφο όμως. Ε, το θύμισαν και το G8 και το G20 φέτος. Κάποιες φορές ε, τέτοιες ενέργειες χρειάζονται και είναι ευπρόσδεκτες. Επίσης, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια της αγοράς, να ξέρουμε ποιος τοποθετείται πού, τι θέση καλύπτει και τι αξιώσεις ή συμβάσεις έχει στην αγορά. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και τη λειτουργία της αγοράς ανάλυση της λειτουργίας της αγοράς είναι κάτι που θα πρέπει πάντοτε να ζητούμε να γίνεται και να προωθούμε οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. Το φαινόμενο λοιπόν της έντονης διακύμανσης των τιμών είναι κάτι που δεν θέλω να αναλύσω περαιτέρω εδώ. Απλώς να πω ότι υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν γίνει και για τα αίτια και για τα αποτελέσματα της κρίσης του 2008. Ένα από αυτά, από την, μία από αυτές μάλλον από την Ήπρη, είναι ιδιαίτερα διεξοδική. Το άλλο σημείο που ήθελα να σχολιάσω είναι ένα-δυο ζητήματα που αφορούν το τι λεπτομερώς θα κάνει από εδώ και μπρος η Επιτροπή. Πολύ συγκεκριμένα, το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του, αφού εξέτασε την ανακοίνωση πέρυσι το Μάιο, ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή το επεξεργαζόμαστε και θα φροντίσουμε να έχουμε χειροπιαστές προτάσεις για το πώς να μεταφράσουμε τις γενικές πολιτικές μας κατευθύνσεις, τις ανακοίνωσες δηλαδή, σε δράσεις. Το φύλλο, τα θέματα των φύλων είναι θέματα στα οποία όντως δεν προσδώσαμε ιδιαίτερη προσοχή, αλήθεια είναι αυτό. Είναι σημαντικός ο ρόλος των γυναικών, ε, ίσως δόθηκε και κάποια προσοχή, αλλά όχι αρκετή. Και είναι πολύ σημαντικός ε, ο τύπος γεωργίας, το είδος γεωργίας που προωθούν οι γυναίκες. Ή μάλλον η σχέση είδους καλλιέργειας με το ρόλο των γυναικών και με τον ρόλο των γυναικών στη γεωργία καθώς και το τι καθήκοντα λαμβάνουν ε, για τη διατροφή της οικογένειας και σε οικογενειακό επίπεδο. Τώρα για την πολιτική συνοχή μας, για την ανάπτυξη. Έτοιμα της κυρίας Κέλλερ σχετικά. Η κοινή αγροτική πολιτική μας απασχολεί από τη σκοπιά της μελλοντικής της μεταρρύθμισης και από τη σκοπιά της ανάπτυξης. Όλα αυτά βρίσκονται σε διαβουλεύσεις. Όμως θα πρέπει να λάβουμε τις αναπτυξιακές διαστάσεις υπόψη και στη μελέτη αντικτύπου που έχει ήδη ανατεθεί και διενεργείται θα δούμε, θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι από το θέμα των εξαγωγικών επιδοτήσεων και μόνον να δούμε τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν στις αλλαγές των τιμών διεθνώς λόγου χάρη. Στον αγώνα αυτών των τιμών υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι βεβαίως. Τώρα θα ήθελα να σταματήσω εδώ τα σχόλιά μου και ο συνάδελφος από την Γενική Διεθνή ΕΚΟ θα κάνει τα σχόλια για τις υπόλοιπες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε. Κύριε Κόρτες Λάστρα, ζητήστε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στην κυρία Τσίμερ για την έκθεσή τη. Πιστεύω ότι είναι μια πλήρης έκθεση. Και μάλιστα μας έρχεται σε μια στιγμή σημαντική. Στηρίζω απόλυτα λοιπόν τα λόγια του κυρίου Νέσερ που λέει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται κερδοσκοπία όσον αφορά τα επισητιστικά και είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, κάνει, να κάνουν ό,τι μπορούν. Ακούσαμε για τους ανθρώπους που δεν έχουν αφάνει στον κόσμο, ξέρουμε ότι το νούμερο όλο και αυξάνεται Ξέρουμε τι γίνεται με τις τιμές των τροφίμων που αυξάνονται μερικές φορές. Ξέρουμε ο κόσμος ζει στην Ήπεθρο και υποφέρει από την κερδοσκοπία αυτή στα αγροτικά προϊόντα. Έχω ένα πολιτικό στόχο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ και που θα έπρεπε να τον αναλάβουμε όλοι. Είναι κάτι γενικό. Θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε τρία τμήματα. Πρώτα απ' όλα, συμμαχία για την επιστημική ασφάλεια και τη διατροφή του κόσμου. Δεύτερον, στήριξη στη μεταρρύθμιση του ΦΑΟ. Και τρίτον, να υπάρξει χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά τα επιστημιστικά ζητήματα στον κόσμο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Κίγκαν πάκλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ναι, αλλάξαμε θέσεις εδώ είμαι τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά για την πολιτική μας επιστηστικής βοήθειας και όσον αφορά επίσης και την σύμβαση για την επιστηστική βοήθεια. Θα συμπληρώσω βασικά αυτό που εξήγησε και ο συνάδελφος. Όπως θα ξέρετε, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια της Επιτροπής, η επιστηστική βοήθεια και η διατροφή είναι ο μεγαλύτερος τομέας, το μεγαλύτερο τμήμα είναι ένα τρίτο με 40% του συνόλου. Συνεπώς για μας ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες ότι η επισητιστική αυτή βοήθεια να προσφέρεται πιο αποτελεσματικά και να είναι πιο αποδοτική. Πέρυσι λοιπόν είχαμε μία ανακοίνωση όσον αφορά την ανθρωπιστική επιστηστική βοήθεια με κύριο στόχο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο αποδοτικοί όσον αφορά την ε, βοήθειά μας αυτή. Να προσφέρουμε δηλαδή την καλύτερη δυνατόν βοήθεια ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί, στηρίζοντα του πιο ευάλωτου πληθυσμού που κινδυνεύουν από ανθρωπιστική κρίση ή που βρίσκονται σε ανθρωπιστική κρίση. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε λιγάκι την απάντηση που δίνουμε σε ανθρωπιστικές κρίσεις και να αλλάξουμε λίγο την αντίδρασή μας που ήταν απλώς διανομή τροφίμων και να δούμε μήπως υπάρχουν και άλλα μέσα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Οπότε πολιτική επισητιστικής βοήθειας προωθεί την χρήση και άλλων μέσων βάτσας ε, ή άλλων περιπτώσεων που μπορούν να βοηθήσουν στην περίπτωση ε, επισητιστικής ε, κρίσης πέρα από τη διανομή δηλαδή αλευρίου, ριζού κτλ. Οι δύο ανακοινώσει λοιπόν που είχαμε προχώρησαν, παρακολουθήσαμε πολύ καλά την κατάσταση και κάθε φορά που ήταν αυτό δυνατό προσπαθήσαμε από την αρχή που είχαμε μια επίγουσα κατάσταση να προσφέρουμε και μια παρέμβαση πιο μακροπρόθεσμα επισητιστικής αρρωγής. Βέβαια δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό πάντα γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανθρωπιστική ε, βοήθεια και την ανάπτυξη. Το πρώτο βασίζεται καθαρά σε ανθρωπιστικές αρχές, ενώ η αναπτυξιακή βοήθεια βασίζεται σε άλλες αρχές, στο δικαίωμα, ε, στα τρόφιμα και άλλα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Κάτι άλλο τώρα που αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωσή μας είναι διατομειακές αποφάσεις όσον αφορά τη διατροφή. Πολλές φορές οι γυναίκες και τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από επισητιστικές κρίσεις και είναι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί. Τώρα, συγχρόνω με αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε όσον αφορά την ανθρωπιστική επισητιστική βοήθεια που θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματική, Κάνουμε και προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυγχρονίσουμε την ε, σύμβαση για την επισητιστική βοήθεια. Είναι του 1999 και πρόκειται για ένα παλιωμοδίτικο μηχανισμό που έχουμε στη διάθεσή μας και που είχε να κάνει με το πώς θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε τα αποθέματα που είχαμε από τη δεκαετία του 60. Οπότε, προκειμένου να μπορέσουμε να πιέσουμε και να προωθήσουμε την ιδέα και τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει τώρα ηγετικό ρόλο προκειμένου να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για να τροποποιηθεί η σύμβαση αυτή. 14 Δεκεμβρίου του 2010 μάλιστα τελικά Επίσημα ε, δεχτήκαν όλα τα μέλη την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης και οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν αμέσως. Τώρα είμαστε σε πολύ εντατική περίοδο διαπραγματεύσεων. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζουμε ώστε να έχουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα βάσει το οποίου ιδεοδός θα συμφωνήσουμε επί της βάσης του περιεχομένου της σύμβασης όταν θα εκπνεύσει η τρέχουσα σύμβαση που είναι τέλη Ιουνίου του 2011. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κυρία Στίφλερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κι εγώ. Με συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στην εισηγήτρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 31 Οκτωβρίου μάλλον 31 Μαρτίου 2010, ανέκρινε δύο ανακοινώσεις. Η μία για την επιστημιστική βοήθεια και μια άλλη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, ακριβώς επειδή η επίγουσα βοήθεια, η αποκατάσταση και η ανάπτυξη είναι άρρηκτα στεδεμένα μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, η πρόοδος που επιτυχάνεται είναι πολύ διαφορετική, ανάλογα και με την πολιτική δέσμευση που διαπιστώνεται. Η η επίγουσα βοήθεια γίνεται βάσει ειδικών κριτηρίων και υπάρχει και πλήρης αξιολόγηση, έτσι δεν είναι. Ο συντονισμός τώρα των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των αναπτυξιακών οργανώσεων επιτόπου και ο συντονισμός με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κράτων μελών είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί. Γιατί από τη σύνδεση όλων αυτών μεταξύ τους μπορεί να πετύχει και η επισητιστική βοήθεια. Πρέπει λοιπόν να το φροντίσουμε αυτό. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να μπερδευόμαστε και να μην είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Η συγκήτρια για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, παρακαλώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τις πολλές προτάσεις που ακούσαμε στη συζήτηση και που θα είναι χρησιμότατες κατά την επεξεργασία της έκθεσης Τονίζω και πάλι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεργαστώ με τους σκιώδεις εισηγητές των διαφόρων ομάδων, ώστε να μην χάσουμε μια ευκαιρία εδώ να παρουσιαστούμε ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο μετά με τρόπο σωστό απέναντι σε αυτή την προβληματική. Θέλαμε η Επιτροπή να αναλάβει μια τέτοια έκθεση και ένας βουλευτής είπε ότι αυτή η έκθεση έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Υπάρχουν και προσδοκίες προς εμάς το Κοινοβούλιο. Αφενός να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να αναλύσουμε σωστά την κατάσταση και να καταδείξουμε προοπτικές. Να αναφέρομαι τις προσδοκίες που, και τις απαιτήσεις που έχουμε προς τα θεσμικά όργανα. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια έκθεση υπόκειται και αυτή σε σαφείς κανόνες εις ό,τι αφορά το εύρος της. Και τονίζω από τώρα ότι είναι πολύ σημαντικό από κοινού να κάνουμε διευκρινήσεις, να επιφέρουμε βελτιώσεις μέσα από τις τροπολογίες, ούτως ώστε να είμαστε ακριβέστατοι. Τίποτε δεν είναι χειρότερο σήμερα από το να έχουμε σε τελευταία ανάλυση μια γενικόλογη έκθεση που χάνεται μέσα στις κοινοτοπίες. Έτσι δεν θα έχουμε συμβάλει όπως πρέπει σήμερα. Να πω στην Κομισιόν ότι βεβαίως και ενδιαφέρομαι να ενημερωθώ για την πορεία των εργασιών ε, επί του εγγράφου υλοποίησης που αναφέρατε, γιατί το Συμβούλιο ανέθεσε στην Κομισιόν να προετοιμάσει ένα τέτοιο έγγραφο ε, υλοποίησης. Θα ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε και εμείς τις σχετικές πληροφορίες και να παρακολουθήσουμε και εμείς ε, αυτή τη διαδικασία, να είμαστε συνδεδεμένοι μαζί σας για να μπορέσουμε να βρούμε και τις σωστές προτεραιότητες. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι στην Κομισιόν και στις ειδικέ επιτροπές υπάρχει η τεχνογνωσία ούτω ώστε να παρακολουθούνται οι συζητήσεις και να γίνεται η σωστή επεξεργασία των θεμάτων. Και όταν εγώ καταπιάστηκα με την έκθεση αυτή, διαπίστωσα ότι το θέμα της διακύμανσης των τιμών στην αρχή έπαιξε ρόλο ε, το είδα αυτό για την ε, κρίση, αλλά στην αρχή δεν είχα καταλάβει πόσο πολύ σημαντικό ήταν αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να αλλάζουμε τις προτεραιότητές μας μετά μέσα από την ενημέρωση, την καλύτερη ενημέρωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συμβάλλει εδώ με χρήσιμο τρόπο η έκθεση. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, γεωργική μεταρρύθμιση, είναι σημαντικό ως Επιτροπή Ανάπτυξης να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και παραπέμπω σε μια συζήτηση που εμείς είχαμε κάνει μεταξύ των συντονιστών για το αν χρειάζεται να γνωμοδοτήσουμε ως Επιτροπή Ανάπτυξης για την ΚΑΠ. Θα ήταν τεράστιο πρόβλημα αν δεν το είχαμε κάνει Πολύ καλά κάναμε και αποφασίσαμε υπέρ της γνωμοδότησης, ε, διότι εδώ το αίτημα είναι να έχουμε συνεκτικές πολιτικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και νομίζω επίσης ότι κατά τη συζήτηση αυτή για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν πρέπει να υποτιμούμε ένα πράγμα. Ε, Εκπήρας λέω ότι είναι πιθανό στα διάφορα κράτη-μέλη και με τους γεωργούς να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Οι γεωργοί καταλαβαίνουν πολύ καλά τα θέματα και ξέρουν τις βασικές προϋποθέσεις για την παραγωγή τροφίμων, ε, εντοπίζουν τις ελλείψεις ή τους περιορισμούς ε, επουδενή οι ε, συνεταιρισμοί, οι ενώσεις των παραγωγών στην Ευρώπη ε, που δεν είδε ισχύει ότι δεν κατανοούν τα προβλήματα με την, ε, τις τιμές, ε, την υπερπαραγωγή και βεβαίως ξέρουν ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν στην Ευρώπη. Άρα μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση μαζί τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Καλό θα ήταν να το συμπεριλάβουμε. Επίσης κατάλαβα κάτι που νομίζω σχεδόν όλοι το είπατε να πούμε δηλαδή για την κατάσταση των μικρών γεωργών, το παραγωγικό τους δυναμικό, την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη και θέση στις χώρες τους και το ρόλο τους στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να το αναδείξουμε σε ένα κύριο θέμα στην έκθεση. Πολλά προβλήματα έχουμε, αλλά σε τελευταία ανάλυση ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα στηρίζεται και θα προσανατολίζεται προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εφαρμόζεται μαζί με τη βοήθεια των ανθρώπων. Όλοι μαζί θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Επίσης, τέλος, μια παρατήρηση ακόμη Καλό θα ήταν, πιστεύω, αν με σαφέστερο τρόπο από ό,τι μέχρι τώρα και μέσω των ανακοινώσεων ε, της Κομισιόν και μέσα από το δικό μου έγγραφο εργασίας, αναδεικνύαμε καλύτερα το θέμα της ευθύνης μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα με την δική μας στρατηγική για την αηφορία και τη βιωσιμότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν η εργασία μας αυτή να συνδεθεί με το γενικότερο θέμα της στρατηγικής βιωσιμότητας ή αηφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς θα ε, πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρος. Επαναρχόμαστε στην ημερήσια διάταξη για την προβληματική των ε, κατεξοδότηση πράξεων και το δημοκρατικό έλεγχο των ε, μηχανισμών στήριξης. Κύριε Γκέρενς, έχετε το λόγο για τα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, τα έχουμε πει λίγο πολύ όλα. Αλλά ακόμα και έτσι δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι τα έχουν καταλάβει όλοι όλα. Κοιτάξτε, είναι η ιστορία των δύο νομοθετικών ε, πτυχών. Το Συμβούλιο δεν κουνάει καθόλου από τη θέση του. Από τότε που ανέλαβα εγώ αυτή την ε, έκθεση, έκανα τα πάντα για να μπορέσω να επιταχύνω τα διάφορα μέτρα όσον αφορά την μπανάνα και να ξέρετε ότι πολλές φορές κερδίσαμε. Ιδιαίτερα όσον αφορά την προνομιούχα ε, θέση των ε, παραγωγών. Αλλά εκεί που κολλάει το πράγμα είναι στην έγκριση των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Προσπάθησα και στην Κισάσα να εξηγήσω την ε, θέση μας. Και ήμασταν οι μόνοι που τους εξηγήσαμε περί τίνος πρόκειται. Πρέπει επίσης να σας πω ότι οι συνομιλητές μας από την πλευρά των χωρών και δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Να ξέρετε ότι έχουν μια πολύ λαθασμένη εντύπωση για τη δουλειά μας εδώ και για την θέση της δικιάς μας Επιτροπής. Εγώ προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι κάναμε τα πάντα για να τους ικανοποιήσουμε όσον αφορά τις διεκδικήσεις τους. Μία από τις μεγάλες τους ανησυχίες καθησυχάστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό. Και ποια ήταν αυτή η ανησυχία τους ήταν ότι η καθυστέρηση όσον αφορά την εκταμίευση του πρώτου τμήματος των 180 ε, δις, η καθυστέρηση αυτή ε, μπορεί να οφείλεται σε μια πλήρη απώλεια του πρώτου τμήματος. Αυτό, αυτή ήταν η ανησυχία τους. Εγώ τους καθησύχασα και τους εξήγησα ότι περίπου ομόφωνα το Κοινοβούλιο ε, προσπαθεί να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Ακόμα κι αν δεν πληρωθούν γρήγορα. Συνεπώς, εδώ υπάρχει και μια δουλειά απειθούς που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους ε, εταίρους μας από τις χώρες ΑΚΕ. Αυτό που εμένα με σοκάρει σε αυτή την υπόθεση είναι ότι όσον αφορά τα κοινοβουλευτικά προνόμια, εδώ βρισκόμαστε σε ευθύνουσα πορεία. Ξέρετε τα δικαιώματά μα όσον αφορά την επιτροπολογία. Στην προηγούμενη θητεία μου είπαν, εγώ δεν ήμουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε, στην προηγούμενη θητεία, αλλά μου εξήγησαν ότι για 10 περίπου πράξεις το Κοινοβούλιο ε, καμιά δεκαριά φορές ε, ζήτησε κάτι. Και 10 φορές χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξανακάνει τη δουλειά. και δεν ε, πετύχαμε. Στις προτάσεις πάντως που κάνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή, είμαστε ακόμα πιο πίσω σε σχέση με τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προηγούμενη θητεία. Ενώ η συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 290, έτσι όπως εμείς το καταλαβαίνουμε, μας δίνει σαφή δικαιώματα για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε τέτοιες περιπτώσεις. Και το κοινοβούλιο μας, τουλάχιστον εμείς έτσι το καταλαβαίνουμε, δεν θα πρέπει να βρίσκει εμπόδια. Και δεν πρέπει να μας ε, ξεγελάνε και να γυρνάμε γύρω-γύρω χωρίς αποτέλεσμα. Πρέπει να έχουμε λόγο. Αυτά λοιπόν για να διευκρινίσω τις θέσεις μας. Δεν μπόρεσα να είμαι παρόν εδώ όταν ο Γκί Μίτσελ παρουσίασε τη γενική θέση της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου μας για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν ικανοποιητική η απάντηση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ απευθύνομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της λέω το εξής. Ξέρετε ότι πολλοί από εμά σας στηρίζουμε σε αυτά που θέλετε να πετύχετε όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και την αναπτυξιακή βοήθεια. Και σας στηρίζουμε ακόμα και εκεί που δεν έχετε δικαίωμα λόγου για την εξωτερική υπηρεσία. Ξέρω ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δύσκολη. Και εδώ δεν θέλω να μου απαντήσετε, γιατί θα μπορούσε να σας φέρει σε δύσκολη θέση. Όχι. Αλλά εδώ τι λέμε. Είχαμε εδώ τη Lady Άστον, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν μας απάντησε ικανοποιητικά. Θα επανέλθουμε σε αυτό στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Το Συμβούλιο από την πλευρά του δεν ήταν καν παρόν στην Κινσάσα. Αυτή φαίνεται είναι η νέα λογική της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Το Συμβούλιο λοιπόν δεν ήταν παρόν, το Συμβούλιο το οποίο θέλει να καταπατήσει τα κοινοβουλευτικά μας προνόμια, τα δικαιώματά μας, αλλά δεν έρχεται καν να μιλήσει μαζί μας. Είναι θλιβερό πιστεύω να μην έχουμε διάλογο με το Συμβούλιο. Δεν έχουμε καν τα μέσα να του παρουσιάσουμε τις δικές μας απόψεις, τη γνώμη μας σε βάθος. Όχι. Αυτό καταπατάει τα κοινοβουλευτικά δικαιώματά μας. Εμείς Μιλάμε για περισσότερη δημοκρατία σε πολλές χώρες. Ε, δεν είναι με τέτοια παραδείγματα που τους δίνουμε που οι χώρες αυτές θα εμπνευστούν για περισσότερη δημοκρατία. Τώρα, η κατανομή καθηκόντων καταλήγει στο ότι κάποιος πρέπει να αναλάβει το καθήκον αυτό. Και εγώ θα γίνω μουτζούρι. Τι να κάνουμε, θα αναλάβω εγώ αυτή τη δουλειά για τις χώρες ΑΚΕ. Αλλά αν συνεχίσει αυτή η έλλειψη κατανόησης, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξηγήσουμε παρόλα αυτά τη θέση μας. Και υπάρχουν και οι εταίροι μας οι οποίοι θέλουν περισσότερη δημοκρατία και τους συμφέρει οι εταίροι τους από τις χώρες Κοτονού να μην έχουν πιο αποδεινωμένη θέση καθ' άλλου. Στις διαπραγματεύσεις λοιπόν που δεν γίνονται, εξαιτία Επιτροπής και του Συμβουλίου, δυσκολεύουν την κατάσταση. Η τελευταία λέξη όμω δεν έχει υποθεί ακόμα. Στην επόμενη Ολομέλεια, από ό,τι έχω καταλάβει, θα μπορέσουμε να πούμε τη γνώμη μας. Και έτσι φιλοδοξώ να περάσουν οι θέσεις του Κοινοβουλίου έτσι όπως εγκρίθηκαν αυτές τον Νοέμβριο. να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, αλλά όχι τα ουσιώδη. Γιατί υπάρχει ένα όριο. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε κάτω από αυτό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και με κάθε σεβασμό που έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω ειλικρινά ότι κάνετε λάθος. Και ότι αν δεν κάνετε εσείς μια χειρονομία προς το μέρος μας, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εδώ εμείς έχουμε παίξει το δικό μας ρόλο. Το άρθρο 290 της Αθήκης της Λισαβόνας το ερμηνεύουμε όπως το ερμηνεύουμε εμείς και επιμένουμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιμένει σε αυτό. Και ορισμός, μάλλον, συγγνώμη, και η θέση που στηρίζω εδώ δεν είναι δικιά μου προσωπική, πια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι καν η θέση της κοινοβουλευτική αυτής επιτροπής. Όχι, είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολόκληρου. Είναι ξεκάθαρο. Και σε αυτή τη βάση θα ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, έχετε το λόγο κύριε Τιελάν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρενς για το εξαιρετικό έργο που έκανε με αυτή την έκθεση. Εδώ πρέπει να καλύψουμε τις προσδοκίες των παραγωγών μπανάνας των χωρών με τους οποίους συνεργαστήκαμε και είχαμε και συζητήσεις και τους λάβαμε υπόψη μας στην πρώτη ανάγνωση του κειμένου. Όπως έχει υποθεί προηγουμένως, αυτό που έχουμε να κάνουμε σε αυτές τις δύο διαδικασίες ανάγνωσης είναι να δούμε τα διαθεσμικά ζητήματα πέραν μίας τροπολογίας, όλα, όλες οι άλλες έχουν να κάνουν με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις που μας απασχολούν εδώ και μήνες. Για τις μελλοντικές λοιπόν αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε παρανόηση ε, και ιδίως ως προς τους ε, ομολόγους μας των χωρών και. Εδώ έχουμε έρθει πραγματικά σε δύσκολη θέση. Διότι αφού νομίμως έχουμε λάβει το δικαίωμα να προβλέψουμε συνοδευτικά μέτρα από την Επιτροπή. Τελικά, οι ομόλογοι μας των χωρών ΑΚΕ δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ που να γεμίσει τα ταμεία τους ε, για την μπανάνα, όπως προβλέπουν οι συμφωνίες της Γενέβης. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε για τους ομολόγους μας της ΑΚΕ, όσα προέβλεψε η τελευταία συνάντηση, η μεικτή συνάντηση βουλευτών στην Κινσάσα, ε, όπου υπό την πρωταβουλία του κυρίου Γκέρενς συζητήσαμε την, ε, το κατά πόσο είναι βάση η προσέγγισή μας. Έτσι λοιπόν σήμερα επαναλαμβάνουμε αυτήν την έκκληση. Εδώ και χρόνια είμαστε αποτελεσματικοί εταίροι, προκειμένου λοιπόν να διασυνδέσουμε περισσότερο τις δικές τους διεκδικήσεις με το τι γίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ενεργήσουμε τα ερχόμενα χρόνια για τη σωστή χρήση των πόρων της εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην παγιδευτούμε εμείς οι ίδιοι. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να κατανοήσουν ότι επιτέλους πρέπει η διαφάνεια να βρίσκεται στην καρδιά της δράσης μας και της λήψης των αποφάσεων αυτό είναι το πνεύμα της συνθήκης και της ίδιας της ιστορίας. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα η Επιτροπή με τον κύριο Ντομένη Κοντερόσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά όσα είπε προηγουμένως ο κύριος Μίτσελ και έπειτα και όσα είπε ο κύριος Γκέρενς. Θα ήθελα εδώ να εξηγήσω κάποια πράγματα που νομίζω ότι προκάλεσαν παρανοήσεις. Πρώτα απ' όλα δεν παίρνει το μέρος του ενός του άλλου θεσμικού οργάνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μας θέση είναι ότι υπερασπιζόμαστε συλλογικά συμφέροντα, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής καθεαυτής, είτε ενδεχομένω των εταίρων μας από τις χώρες ΑΚΕ. Αυτό θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια της ε, συνθήκης της Λισαβόνης και, Λισαβόνας και των πρωτοβουλειών και αρμοδιοτήτων προβλέπουν που προβλέπονται μάλλον για τα διάφορα θεσμικά όργανα. Εμείς λοιπόν εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της διοικητικής απλούστευσης. Και σε καμία περίπτωση για τον αντίθετο σκοπό για να επανέλθουμε στην μπανάνα. Εδώ μιλάμε για εφαρμογή μέτρων εντός τριετίας. Όπως λέει το στατικικό έγγραφο υπάρχει προβλεπόμενη ανάλυση. Η Επιτροπή όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα αυτό για τις κατατοξιοδότηση πράξης, έθεσε επιτάπητος μία πρόταση, η οποία στοχεύει να ενισχύσει τι αρμοδιότητε και το δημοκρατικό έλεγχο που ήδη προβλεπόταν. Αναγνωρίζουμε λοιπόν, όσα ήδη είπε ο κ. Γκέρεν, ότι πέρυσι για τα έγγραφα αυτά τα στατηγικά, όπου υπήρξε και το ζήτημα, ίσως δεν ήταν πλήρης η διαδικασία, ίσως έπρεπε να γίνουν κι άλλα. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να ε, διευκολύνουμε τα πράγματα. Προτείναμε μια διαδικασία που δίνει πολύ περισσότερα δικαιώματα και εξουσίε για να το πω έτσι, στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να αναγνωριστούν οι τροποποιημένε πλέον αρμοδιότητέ του και οι επιθυμίε του, οι προσδοκίε του όταν τα συζητήσαμε και στο επίπεδο των στρατηγικών εγγράφων. Ιδίω με την ευκαιρία τη μπανάνα. Το άλλο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι στην τροποποίηση του κανονισμού Ήδη ο κανονισμός ορίζει ποιες είναι οι χώρες, ποια τα κριτήρια για την απονομή πόρων. Ορίζει στόχους. Ορίζει τι πρέπει να περιέχουν τα έγγραφα πολιετούς στρατηγικής τεκμηρίωση, αξιολόγηση, εξετάσεις και μελέτες. Εφόσον πρόσφατα εγκρίθηκε το κανονισμός για την επιτροπολογία, το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου, scrutiny right, του Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου, όλα αυτά διαφυλάσσονται. Το να κατηγορούμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο δεν θέλει να σεβαστεί τη συνθήκη της Λισαβόνας ή ότι παίρνει τη θέση, συμπαρατάσσεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, νομίζω ότι αυτό δεν ε, αρμόζει εδώ. Νομίζω ότι ως τώρα πραγματικά υπήρξαμε οι καλύτεροι δημοσιολαβητές. Προσπαθήσαμε μάλιστα να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, διότι συμφωνούμε όλοι, είναι υψηλό το ποσό, 90 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να το αγγίξουμε. Θα υπάρχει όμως ένα πρόβλημα υλοποίησης, διότι θα πρέπει να συμπιεστεί η υλοποίηση εντό μιας τριετίας και να σεβαστούμε και τους κανόνες που αποφασίστηκαν ακριβώς από αυτό το κοινοβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ναι, ένα πρόβλημα με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει όμως με την επόμενη ευκαιρία, με το έγγραφο πλαίσιο με το έγγραφο μάλλον για το δημοσιονομικό πλαίσιο, τότε να δούμε ποιε ακριβώ θα είναι οι κατεξουσιοδότηση πράξει. Ωστότε, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε και τη δυτική χρήση των όσων προβλέπει αυτό το έγγραφο. Δηλαδή τα όσα θα συμπεριλαμβάνει το στατηγικό έγγραφο και όσα δεν θα είναι κατεξουσιοδότηση πράξης. Ε, προσωπική παρατήρηση τώρα αυτή, αλλά μου φαίνεται δύσκολο σε κάποια χώρα τα στρατηγικά έγγραφα να θεωρούνται κατά νομοθετικές μάλλον πράξεις ή ιονί νομοθετικέ και όχι εφαρμοστικές. Θα διερευνήσω το σημείο βέβαια αυτό, πάντως πρόεδρε προσπάθησα να αποσαφηνίσω λίγο τα πράγματα. Δεν θέλω να παραμείνουν αμφισημίε ότι είμαστε με το μέρο του Συμβουλίου, ότι είμαστε με το μέρο του Κοινοβουλίου. Όχι. Θέσαμε επιτάπητο στο πρόβλημα. Δεν αποφύγαμε και τα επικριτικά σχόλια του Συμβουλίου που θεώρησε ότι πηγαίνουμε πολύ μακριά σε σχέση με όσα μπορούσαμε να κάνουμε ή όσα αρχικά είχαμε προτείνει. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Έχοντα υπόψη ότι θα πρέπει να περιμένουμε και τρία χρόνια πριν τον νέο κανονισμό για το μέσω συνεργασία. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Γκέρεν. έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Παρά την καλή σας θέληση, δεν με πείσατε πλήρω. Λυπούμαι εγώ πρώτος. Παρά τη φιλική σχέση που έχουμε, εσείς ως εκπρόσωπος της Κομισιόν με τα μέλη της Επιτροπής μας. Δεν θα υποχωρήσω καθόλου, ούτε σπιθαμή, σε σχέση με όσα είπα. Τώρα, μας είπατε, να, ένα έγγραφο που προβλέπει την κατανομή των 90 εκατομμυρίων στις χώρες που ορίζει το στρατηγικό έγγραφο. Ανακεφαλαιώνω, δεν ακριβώς αυτά τα λόγια σας. Και τι καθυστερήσεις μπορεί να υπάρχουν. Λοιπόν, εάν είναι εντάξει τα στρατηγικά σας έγγραφα, ε, θα έπρεπε να περάσουν αυτομάτως. Δεν θα υπήρχαν αμφισβητήσεις, ούτε θα υψώναμε τη φωνή μας. Αυτό το είδαμε και με άλλα έγγραφα που συζητήθηκαν σε επίπεδο ομάδα εργασίας D, της οποίας προεδρεύω. Ε, προσπαθήσαμε πάντοτε να δείχνουμε κατανόηση απέναντί σας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και όταν προβάλαμε διαφωνίες, ήταν στο κατά πόσον σωστά κατανείμονται οι πόροι, τα κονδύλια, δηλαδή βάσει τη αναπτυξιακή βοήθεια και τη εξωτερική μα πολιτική ω κριτήριο. Εδώ μας είπατε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η κυρία Άστον όμω, που είναι η αντιπρόεδρο και πρόεδρο του Συμβουλίου, θα πρέπει να ασκήσει και λίγο την πυγμή τη, προκειμένου να διατηρήσουν και εκείνη μια πιο σταθερή στάση και να είναι πιο ευνοϊκή. Εδώ δεν μπορώ να προδώσω τη θητεία μου. Δεν μπορώ παρά να πω ότι η κατάσταση σήμερα για μας είναι απαράδεκτη. Γι' αυτό στη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης ξεκινάμε από την αρχή. Εδώ δεν θέλουμε να διαιωνίζουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ε, δεν είναι αυτός ο στόχος μας, να προβάλλουμε εμπόδια. Τώρα, τι θέλουμε, ένα στρατηγικό έγγραφο να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να αλλοιώσει τη βασική νομοθεσία. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το αν θα επιλέξουμε αυτή την κατεύθυνση. Και για να ολοκληρώσω και να διασκεδάσω λίγο από του συναδέλφου, εγώ ίδιο έχω υπάρξει μέλο εκτελεστική εξουσία Και ο ίδιος είχα την προσωπική μου εμπειρία και είδα ότι οι βουλευτές είναι άνθρωποι που μας δυσκολεύουν τη ζωή. Και ξέρω ότι αυτοί που κυβερνούν δυσκολεύονται πάρα πολύ να το κάνουν με τέτοιου συνεργάτε. Όμω. Υπάρχει δυνατότητα συνύπαρξη. Μπορεί το ευρύτερο σκηνικό του αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου να λειτουργεί. Υπάρχουν προποθέσει για να γίνει κάτι τέτοιο. Δώστε μα την ευκαιρία να ασκήσουμε αυτόν τον έλεγχο. Και όλες οι υποψίες που περίπτανται θα ε, εξαλειφθούν στην πράξη. Θα εξατμιστούν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για τις δύο του κ. Μίτσερ και του κ. Γκέρενς για τη δεύτερη ανάγνωση. Απόψε στις 7.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 que je veux soumettre à la Commission aussi longtemps que sa position définitive n'est pas encore arrêtée, ce qui est le rôle même de notre. Η δημοσιονομική στήριξη μιλάει για την εξωτερική χρηματοδότηση σε χώρες εταίρους εφόσον οι χώρες προορισμού τηρούν κάποια κριτήρια. Και εφόσον χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά τελικά υπέρ της βελτίωσης των δημοσιονομικών της ε, χώρας προορισμού. Τώρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγώ ξέρω έναν δωρητή και μια χώρα προορισμού. Όχι πολύ μακριά από εδώ. Ο δωρητής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα που παίρνει τα κονδύλια είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Όταν διαβάζω την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για το χρόνο, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια αυτά, τίθεται πάρα πολλά ερωτήματα. Σε μια χώρα η οποία θεωρητικά και δεν είναι μόνο μία, αυτή είναι και άλλες χώρες στην ίδια κατάσταση, η οποία εφαρμόζει λιτότητα στα δημοσιονομικά της. Εφόσον λοιπόν ήδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα όσον αφορά την χρήση των ε, δημοσιονομικών πόρων, φανταστείτε οι χώρες οι οποίες συνδέονται με τον δωρητή μέσω λιγότερο αυστηρών ε, προδιαγραφών, ε, καταλαβαίνετε πόσο μάλλον εκεί μας δημιουργούνται ερωτήματα. Τώρα, για να είμαι ξεκάθαρος, εγώ θέλω να δίνουμε τη δημοσιονομική στήριξη, αλλά θέλω να περιορίζουμε τις περιπτώσεις, τις προβληματικές με τη διάθεση αυτών των κονδυλίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβλέπει την ε, πάυση. Υπάρχουν ε, όμως και εμπειρίες πάρα πολύ καλές. Παραμένουν όμως τα προβλήματα σε μερικές περιπτώσεις. Ποιες είναι οι πτώσεις τώρα της δημοσιονομικής στήριξης. Τα αποτελέσματα είναι άλλοτε καλά, άλλοτε άσχημα. Με την ε, αξιολόγηση του 2006 που έγινε, Πουρκίνα Φάσο, μαλαουί κλπ, Ρουάντα, Βιετνάμ, που ζήτησε την αξιολόγηση αυτή ο ΣΑ, διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν θετικές ε, επιπτώσεις για την ορθολογική χρήση των ε, δημοσίων δαπανών και για τον τρόπο που χειρίστηκε ε, τα, το δημόσιο χρήμα η κυβέρνηση στην κάθε μία από τις χώρες αυτές. Όμως, σε άλλες περιπτώσεις τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά. Υπάρχουν ε, επιφυλάξεις και όσον αφορά την αξιολόγηση αυτή που έχει να κάνει με τη δοσιονομική στήριξη και πώς αυτή επηρεάζει την υποχώρηση της φτώχειας, τη δημοκρατία κλπ. Έχω και το σημείο 3 στην έκθεσή μου που αναφέρεται στους όρους εισδοχής στην βοήθεια. Πώς επιλέγονται δηλαδή οι δικαιούχοι χώρες. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα κριτήρια δεν είναι πάντα αυστηρά. Υπάρχει δυνατότητα στα πλαίσια του διαλόγου, νομίζω ότι πρόκειται για το άρθρο 61 της Σύμβασης Κοτονού, που προβλέπει ότι μπορούμε να επιταχύνουμε την κίνηση στα πλαίσια μιας δυναμικής χορήγησης βοήθειας. Υπάρχουν προηγούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η... Με τους δικαιούχους στην ΟΝΕ το ίδιο έγινε. Είχαμε την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή, οι προϋποθέσεις δεν έπρεπε να τηρούνται τη στιγμή εισόδου στην ε, ΟΝΕ των χωρών, θυμόσαστε τότε. Οι υποψήφιες χώρες δεν ήταν απαραίτητο να τηρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά έπρεπε να υπάρχει η τάση που θα οδηγούσε στην τήρηση των προϋποθέσεων. Απριόρι δεν λέω ότι είμαι κατά μια τέτοιας προσέγγισης, αλλά ελοχεύουν κίνδυνοι εδώ. Και η ερώτησή μου είναι, μπορούμε να διαχειριστούμε αυτούς τους κινδύνους. Τι γίνεται αν δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα σε μια χώρα δικαιούχο, που τελικά δεν τηρεί τις προϋποθέσεις και δεν είναι σε θέση να ταποκριθεί στα κριτήρια που έχουμε διαπραγματευτεί μαζί τους. Αναρωτιέμαι επίσης και για κάτι άλλο. υπάρχουν ε, διπλωματικές, γεωπολιτικές θεωρήσεις ή ακόμα και προσωπικές σχέσεις που μπορούν να παίξουν εδώ ρόλο και να επηρεάσουν αυτόν που διαπραγματεύεται από την πλευρά μας με τις χώρες δικαιούχους. Μήπως δηλαδή ο γνώμονας είναι υποκειμενικός. Τώρα σε ένα έγγραφο που δημοσιεύθηκε το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι έτοιμη να εφαρμόσει τα του άρθρου 61 παράγραφος 2 της Συμφωνίας ε, Κοτονού και ότι οι δυναμίες που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά των χωρών δικαιούχων δεν εμποδίζουν να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής ε, στήριξης εφόσον υπάρχουν θετικές προϋποθέσεις και ότι η Κομισιόν παρακολουθεί την κατάσταση μαζί με την λόγο χώρα. Αυτή η δυναμική όμως πρέπει να υπάρχει και όσον αφορά τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του Κοινοβουλίου στις διάφορες χώρες. Και θα ήθελα εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δηλαδή, τι βελτιώσεις έχουν διαπιστωθεί όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό το λέω γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα. Εγώ συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις που έγιναν για την Συμφωνία Κοτονού το 2000. Ε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ δυσκολευτήκαμε να κάνουμε τις χώρες ΑΚΕ να δεχτούν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη συμφωνία. Υπήρχε τεράστια επιφύλαξη από την πλευρά τους, ε, τεράστια δισταγμή. Χρειάστηκε να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει πάρα πολύ για να τους κάνουμε να το καταπιούνε. Ενώ είναι προς το συμφέρον και το δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει η ενδογενής ανάπτυξη χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η κοινωνία των πολιτών δεν αρκεί να υπάρχει και ένα χιόνομα, πρέπει να συμμετέχει. Γιατί αυτή αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα. Και έχει πάρα πολύ σημασία αυτό για τις χώρες εταίρους τις υπονάπτυξη χώρες. Ακριβώς επειδή είναι αδύναμο το εκτελεστικό σύστημα εκεί, άρα και το κοινοβουλευτικό. Άρα πρέπει να υπάρχει και αυτό για να είναι αξιόπιστο το δημοσιονομικό εγχείρημα. Αν τώρα στην δυναμική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχουν και τα δύο, τότε η δημοσιονομική στήριξη κινδυνεύει δεν θα πετύχει τους στόχους της που είναι ιδιαίτερα ευγενείς, αλλά κινδυνεύουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοια προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Κάτι άλλο τώρα που είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι αποφασιστική σημασία, τι είναι το αποφασιστικό και ποιος αποφασίζει για το ότι το σημείο εκκίνησης είναι επαρκές. Δηλαδή ότι οι συνθήκε που επικρατούν σε μια χώρα είναι ικανοποιητικέ. Υπάρχουν και άλλοι δωρητέ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η, η Παγκόσμια συγγνώμη, Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούν τα ίδια κριτήρια ως σημείο κίνησης για να βοηθήσουν μια χώρα. Και ποια είναι τα κριτήρια, η διακυβέρνηση, αλλά μήπως είναι διαφορετική και διαφορετικά τα κριτήρια για αυτήν στη μία περίπτωση και στην άλλη, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Έπειτα, η διαχείριση των δημοσίων πόρων δεν μπορεί παρά να είναι μία. Έτσι. Άρα, δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια. Οι δαπάνε με έναν τρόπο γίνονται. Δεν μπορεί ένα να κάνει το ένα και ένα να κάνει το άλλο. Η διαχείριση είναι μία. Συγκεκριμένη. Πώς τοποθετήσετε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, όταν η δικιά σας άποψη διαφέρει από την άποψη του Διεθνού Ταμείου ή της Παγκόσμιας Τράπεζας, αν είσαστε εσείς πιο γενναιόδοροι ή εκείνοι πιο γενναιόδοροι. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τη συμπεριφορά της χώρας που θέλουμε να στηρίξουμε. Εντάξει, δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες, δεν σας τα πω όλα γιατί θα φάω πάρα πολύ χρόνο. Πάντως, θα ήθελα να με στηρίξει η Επιτροπή μας για να διευκρινιστούν τα εξή. Γιατί έχω τα εξή ερωτήματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο πρώτος δωρητή, ο κύριο δωρητή, είναι σε θέση να επηρεάσει άλλους χρηματοδότες. την Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα, ή το ε, Διεθνές Πιστατικό Ταμείο. Δεύτερον, ποιες είναι οι αντισταθμίσεις για τις χώρες που δεν εποφελούνται από δημοσιονομική στήριξη. Και να σας πω τι εννοώ εδώ. Θα θυμόσαστε όλοι συμφωνία του Ντόνιγκελς που επέτρεψε να διαγραφούν 50 δισεκατομμύρια από την Παγκόσμια Τράπεζα. Έτσι, 50 δισεκατομμύρια χρέος ξαφανίστηκε. Όλες οι χώρες μας συμμετέχουν στην ε, επαναχρηματοδότηση των 50 δισεκατομμυρίων αυτών, χρέος το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν επρόκειτο ποτέ να επιστραφεί. Άρα πρόκειται εδώ πέρα για απλή διαπίστωση που κάναμε και πήραμε αυτή την απόφαση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ιδιαίτερα επέμειναν για πιο αυστηρέ προϋποθέσεις όσον αφορά την διακυβέρνηση και του ίδιου πόρου. Τώρα, υπάρχουν διάφορες χώρες που έχουν δημοσιονομική στήριξη και άλλε που δεν επωφελούνται από δημοσιονομική στήριξη. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις χώρες που δεν έχουν δημοσιονομική στήριξη. Και γιατί, επειδή φταίει η διακυβέρνηση εκεί. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αυτές που τελικά έχουν ακόμα περισσότερο ανάγκη από τα λεφτά αυτά. Δεν είναι αντίφαση αυτό. Θα έπρεπε εδώ να βρούμε μια λύση. Εσείς στις σχέσεις που έχετε με τους εταίρους Διαπιστώνεται αυτή την πρακτική ότι δηλαδή δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο οι χώρες εκείνες οι οποίες δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για δημοσιονομική στήριξη. Πώς θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε. Άλλη ερώτηση κατά τη διακοπή της δημοσιονομικής στήριξης σε μια χώρα. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της απόφασης αυτής στην περιφερειακή ενοποίηση. Και τι εννοώ εδώ. Ας δούμε. Ακτήλε Φαντοστού, παράδειγμα. Αν η Ακτήλε φαντοστού ήταν δικαιούχος δημοσιονομικής στήριξης με αυτά που συμβαίνουν σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να σταματήσει την δημοσιονομική στήριξη. Αλλά τότε θα επλήγεται ολόκληρη η περιοχή. Δηλαδή και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ακτή ελεφαντοστούκη που μπορεί να είναι πιο φτωχή ακόμα. Το γεγονός δηλαδή ότι τιμωρούμε κατά κάποιο τρόπο διακόπτοντας τη δημοσιονομική στήριξη μια χώρα επειδή δεν συμπεριφέρεται καλά έχει επιπτώσεις στην ε, γύρω περιοχή και τι επιπτώσεις τις λαμβάνεται υπόψη. Και τέλος, η δημοσιονομική στήριξη είναι το καλύτερο κίνητρο για την ενδογενή ανάπτυξη. Σας έχω ήδη πει τις σκέψεις μου, αλλά θα ήθελα να ξέρω και ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γι' αυτό. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το εγγραφό είναι επικριτικό. Η δικιά μου η προσωπική θέση, αν θέλετε, είναι πιο ισορροπημένη από αυτήν που αναφέρεται στο κείμενο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή κοινοβουλευτική δουλειά και είναι καλό να επικεντρωνόμαστε στα πιο επικριτικά στοιχεία χωρίς όμως να ε, πλήξουμε μια πρακτική η οποία είναι και πολύ θετική συγχρόνως. Ευχαριστούμε. Κύριε Μασάν, για 15 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εισαγωγικά δύο λόγια να σας πω. Πρώτα απ' όλα. Έχουμε ένα έγγραφο στο οποίο συνοψίζουμε επαφές που είχαμε με διάφορους επιρρογνώμονες για το θέμα της πράσινης βίβλου. Όπως επίσης μετά από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Γκέρενς, πιστεύουμε ότι η πράσινη βίβλο είναι ε, αρκετά πλήρη. Και εμείς συνοψίζουμε δύο πράγματα τα οποία δεν είναι αρκετά εκτεταμένα. Το θέμα της επιλογής των χωρών, για παράδειγμα, όπου δεν υπάρχει ανάλυση για το γιατί τα κριτήρια αυτά είναι τα σωστά. Δεύτερον, εμείς θα θέλαμε σε αυτό το επίπεδο αξιολογήσεων, όπως είπατε και εσείς, θα έπρεπε να μιλάμε και για το πώς επηρεάζουν τα συστήματα λογαριασμών και το χρησιμοποιήσει. Έπειτα υπάρχει δυνατότητα ε, όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη. Με ποια με την έννοια ότι διακόπτεται άπαξ και υπάρχει παραβίαση των ε, κριτηρίων. Όπως για παράδειγμα η ε, διαχείριση, η διακυβέρνηση. Και έτσι καταλήγουμε στο ότι οι δωρητές επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες και προδιαγραφές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία κτλ. Ο κίνδυνος βέβαια είναι ότι οι δωρητές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κάθε φορά που σκέφτονται να κόψουν τη δημοσιονομική στήριξη, γιατί μπορεί να πλήττεται έτσι ακόμα περισσότερο η δημοκρατία στη χώρα. Έπειτα έχουμε το ρόλο του πολιτικού διαλόγου και της αιρεσιμότητας και τη σύνδεση με την απόδοση και τα αποτελέσματα της βοήθειας. Όσον αφορά τις δυνατότητες εδώ, η δημοσιονομική στήριξη, κατά τη γνώμη μας, βελτιώνει και τη συνεργασία ανάμεσα στους χρηματοδότες και την χώρα δικαιούχο. Άρα η εταιρική σχέση και συνεργασία βελτιώνεται μεταξύ τους. Δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα, αιρεσιμότητα, να στηρίξει την κυβέρνηση η οποία θα θελήσει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσει. Σε πολλές χώρες έχουμε τέτοια παραδείγματα. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι. Η αιρεσιμότητα αυτή σε πολλές περιπτώσεις, και το αναφέραμε, καταλήγει σε ένα κατάλογο προτιμήσεων που έχουν κάποιοι δωρητές και μπορεί να έχουν να κάνουν γεωπολιτικά συμφέροντα. Και άρα μπορεί να δυσκολέψουν τις διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο για τη λήψη αποφάσεων. Τρίτον, υπάρχει ο κίνδυνο η αιρεσιμότητα αυτή να είναι υπερβολικά φιλόδοξη. Να είναι μεν θετική, αλλά να είναι υπερβολικά φιλόδοξη και άρα να μην είναι ρεαλιστική και άρα να μην μπορούν να επιτευθούν τα όσα ζητάει η αιρεσιμότητα αυτή. Όσον αφορά το τρίτο σημείο που έχει να κάνει τώρα με τους εθνικούς λογαριασμούς, εμείς έχουμε δυνατότητες, δηλαδή η δημοσιονομική στήριξη το έχει δείξει και η πρακτική δηλαδή σε διάφορες χώρες, ενισχύει τους εθνικούς λογαριασμούς της χώρας και γίνεται κοινοβουλευτικό έλεγχος. Άλλη δυνατότητα είναι η δημοσιονομική στήριξη. Μειώνει μερικές φορές τα παράλληλα συστήματα που έχουμε και ενισχύει το σύστημα εθνικού ελέγχου. Ελοχεύουν όμως και κίνδυνοι εδώ. Αυτό που αναφέρθηκε πριν, ότι οι δωρητές δεν συμπεριλαμβάνουν επαρκώς την κοινωνία των πολιτών, ούτε τα κοινοβούλια ή σε ελάχιστο βαθμό. Το έχουμε δει και αυτό σε πολλές χώρες. Ένας άλλος κίνδυνος είναι η στήριξη δημοσιονομική και στους λογαριασμούς να μην ε, δίνονται αναλογικά. Έπειτα, η εξωτερική ζήτηση για εθνικούς λογαριασμούς μερικές φορές υποτιμάει την ε, εθνική ζήτηση, την εσωτερική ζήτηση. Δημιουργεί πίεση μέσα στη χώρα για να γίνεται απόδοση λογαριασμών στην χώρα που δίνει τα χρήματα, πολύ περισσότερο από ότι να είναι υπόλογη και να δίνει λογαριασμούς μέσα στη χώρα, στους πολίτες της χώρας. Έχουμε διαπιστώσει επίσης προσπάθεια αναρμόνισης οριζόντια για την απόδοση λογαριασμών. Και όχι κάθετα. Στην Κάνα, για παράδειγμα, είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, άρα υπάρχει μεγάλη διαφάνεια απέναντι στους πολίτες για τη δημοσιονομική στήριξη. Έρχομαι στο σημείο 4 που έχει να κάνει με το συνδυασμό της δημοσιονομικής ε, στήριξης με άλλη, άλλα μέσα αναπτυξιακής βοήθειας. Και εδώ υπάρχουν δυνατότητες γιατί η συνολική δημοσιονομική στήριξη και η ανατομής δημοσιονομική στήριξη είναι πράγματα συμπληρωματικά μεταξύ τους. Η ανατομία δημοσιονομική στήριξη έχει σαν αποτέλεσμα εγκάρσιες μεταρρυθμίσεις να ανταποκρίνονται καλύτερα στην εξυπηρέτηση του κόσμου, όπω για παράδειγμα στον τομέα της υγείας ή της εκπαίδευσης. Συγχρόνως, η στήριξη με προγράμματα, αρχές ε, που διαχειρίζονται φορολογικά έσοδα, οι άλλες υπηρεσίες ενισχύουν τη δυνατότητα της κάθε χώρας να διαχειριστεί τις δημοσιονομικές της δυνατότητες. Η στήριξη τώρα στην κοινωνία των πολιτών βελτιώνει τη δυνατότητα απόδοσης λογαριασμού της δικαιούχου χώρας. Το πολιτικό πλαίσιο και το δημοσιονομικό πλαίσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για να χειριστούμε θέματα που έχουν να κάνουν με ειδικού τομεί και να αποφύγουμε το κίνδυνο υπερβολικής φόρτωσης του μηχανισμού. Η κίνδυνη εδώ είναι ότι αν συντηρήσουμε την στήριξη με υπερβολικά προγράμματα, οι δωρητές χρησιμοποιούν περισσότερο κάθε τη στήριξη για να μειώσουν τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με την απόδοση λογαριασμών ε, στις δικές τους χώρες. Πολιτικός διάλογος τώρα. Μπορεί να είναι υπερβολικά φιλόδοξος και παραφορτωμένος, αν υπάρχουν υπερβολικά μέσα συνεργασίας. Σημείο 5 που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να κάνει με την ενίσχυση του ελέγχου για να αποφεύγουμε την διαφθορά. Εδώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχος φυσικά και μειώνει ένα τέτοιο κίνδυνο και βελτιώνει την απόδοση λογαριασμών. Η δημοσιονομική στήριξη επίσης αυξάνει και τα κίνητρα για την αποφυγή της διαφθοράς. Μπορεί επίσης να βελτιώσει και την ε, προβολή της διαφθοράς, να εντοπίζεται δηλαδή πολύ πιο εύκολα και σε περισσότερες περιπτώσεις. Η διαφθορά μειώνει τις δυνατότητες του μέσου αυτού επίσης. Και οι πόροι πολλές φορές από την διαφθορά δεν χρησιμοποιούνται σε τοπικό επίπεδο βέβαια. Έπειτα υπάρχει και ένα άλλο σημείο που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό και είναι η σχέση της δημοσιονομικής ε, στήριξης σε περίπτωση που η κατάσταση σε μια χώρα είναι βάλωτη. Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει πάντα με ναι ή με όχι. Έχουμε συζητήσει με ειδικού και έχουμε διαβάσει πολλά και έχουμε διαπιστώσει ότι η δημοσιονομική στήριξη μπορεί να συνεισφέρει στη σταθερότητα και στην αποκατάσταση τη θεσμική και σε περισσότερες ευθύνες από πλευράς ε, των ε, κυβερνήσεων όσον αφορά την διαχείριση των οικονομικών πόρων και στη Ρουάντα και στη Σιέρα Λεόν έγινε αυτό και στο Αφγανιστάν ακόμα. Με την δημοσιονομική στήριξη δουλεύουν καλύτερα από ό,τι με άλλα μέσα. Όμως, εξαιτία του ευάλωτου της κατάστασης υπάρχουν ε, μεγάλοι κίνδυνοι γνωστοί Η κυβερνητική δομή είναι πολύ αδύναμη γι' αυτό. Και η νομιμότητα της κυβέρνησης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Τέλος, η δημοσιονομική στήριξη σχετικά με την ε, ανάπτυξη. Εννοείται ότι είναι κάτι πολύ θετικό. Ενισχύει και την φορολογική μεταρρύθμιση και την ε, δημόσια δίκηση. Ο πολιτικός διάλογος χρησιμοποιείται για περισσότερη διαφάνεια σε χώρες που έχουν ε, πλούτο. Επίσης βοηθάει και τον σχεδιασμό. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η δημοσιονομική στήριξη μπορεί να μειώσει τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για να βρεθούν ήδη πόροι οι δωρητές συγκεντρώνονται στις δημόσιες δαπάνες και όχι τόσο στα έσοδα. Οι εκταμιεύσεις δεν ε, είναι πάντα προβλέψιμες. Και έτσι ποσοτικά μερικές φορές υπάρχουν ε, προβλήματα εκτίμησης και αναμπερδεύεται το ποσοτικό με το ποιοτικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχετε προσέξει ότι τον τελευταίο καιρό δεν έχω πια άσπρο καρτελάκι, αλλά πράσινο καρτελάκι εδώ μπροστά μου. Δεν είναι γιατί άλλαξα πολιτική ομάδα, σας διαβεβαιώ. Εξακολουθώ να ανήκω στην ίδια πολιτική ομάδα. Ούτε έχει αλλάξει η κατάσταση στην Επιτροπή αυτή. Ο κύριος Γκέρενς είναι πάντα παρόν όταν μιλάμε για την συνεργασία και την ανάπτυξη, όπως και τώρα που μιλάμε για τη δημοσιονομική στήριξη. Μίλησε πριν για ένα σταθμό που δεν φτάνουν ποτέ τα τρένα. Ε, το δικό του το τρένο είναι ένα τρένο προαστιακός που περνάει από κοντά από το κάθε μέρος ξανά και ξανά και ξανά με την σοφία του βοηθάει πάρα πολύ την Επιτροπή μας. Είμαι σκιώδης εισηγητής. Είμαι και συνεισηγητής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ για μία έκθεση δημοσιονομικής στήριξης που θα εγκρίνουμε κατά πάσα πιθανότητα τον Μάιο στη Βουδαπέστη. Είναι λοιπόν αυτό ένα θέμα που με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος. Και όπως είπε και ο κύριος Γκέρενς και ο εμπειρογνώμων μας εδώ, η θέση μας είναι θετική απέναντι σε αυτό. Συγχρόνως, μας απασχολούν πολύ κάποιες δυσλειτουργίες του μηχανισμού αυτού. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε περισσότερο για να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που έχει ο μηχανισμός αυτός και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γκέρενς για την έκθεσή του. Σημερίζομαι τις περισσότερες από τις ιδέες που ανέφερε μεταξύ άλλων την διαβάθμιση της δημοσιονομικής στήριξης, την δυναμική που υπάρχει όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ότι πρέπει να διατηρήσουμε το κριτήριο που λέει ότι ο βασικός στόχος είναι η καταπολέμηση της ένδυας και επίσης ότι πρέπει η προβλεψιμότητα της στήριξης να είναι περισσότερο ορατή. Θέλω να υπογραμμίσω κάποια από τα πλεονεκτήματα που νομίζω ότι έχει το μέσο αυτό δημοσιονομικής στήριξης. Πρώτον, ευνοεί την αρχή που λέει ότι οι χώρες και οι πολίτες νιώθουν δικό τους το έργο που γίνεται με τη δημοσιονομική αυτή στήριξη. Μιλάμε για υποχώρηση της ένδυας. Οι ίδιοι είναι κύριοι των προσπαθειών τους. Δεύτερον, οι χώρες δωρητές ή τέλο πάντων οι οργανισμοί δωρητές. Εδώ ο κύριος Γκέρας πολύ καλά αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα, το Εθνικό Μεσοδικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι χώρες, είναι θεσμοί. Όλοι αυτοί όντω πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς την ίδια κατεύθυνση και μαζί να θέτουν τις προτεραιότητες να μην τις καθορίζουν και να τις επιβάλλουν στις χώρες δικαιούχους, αλλά μαζί τους να τις ε, εντοπίζουν. Έπειτα, στην Επιτροπή μας εδώ, πολύ συχνά, έχουμε συζητήσει για το κόστος των συναλλαγών στον τομέα αυτό. Έχουμε συζητήσει και έχουμε εγκρίνει στην Επιτροπή μας διάφορα κείμενα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, της στήριξης. Και πάντα λέγαμε ότι ο κατακαιρματισμός της στήριξης είναι σε βάρος του στόχου μας. Τέλος, κάποιες συστάσεις για τα επόμενα στάδια της έκθεσης αυτής. Θα μπορούσαμε να τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσουμε τα συστήματα ε, δημόσιας διαχείρισης των χωρών δικαιούχων με στόχο να βελτιώσουν την απόδοση λογαριασμών και τη διαφάνεια. Ακριβώς εδώ ο κύριος Γκέρενς ρώτησε κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έθεσε για ένα προβληματισμό δικό του. Λέει το σύστημα απόδοσης λογαριασμών θα έπρεπε να είναι ενιαίο. Θα έπρεπε να είναι ένα ενιαίο σύστημα για την επιλεξιμότητα πρώτα απ' όλα, για την ε, παροχή της δημοσιονομικής στήριξης αλλά και για την απόδοση λογαριασμών. Δηλαδή να μην υπάρχουν διαφορετικά σενάρια. Να γίνεται άλλη δουλειά για την Παγκόσμια Τράπεζα, άλλη για το Διεθνέ Προστατικό Τομείο, άλλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλη για άλλε χώρε νωρίτε. Όχι. Τη στιγμή που οι περισσότερε από τι χώρε δικαιούχου έχουν δύναμη διοίκηση και του είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό. Θα χάνανε φοβερή ενέργεια για κάτι θα μπορούσε να λυθεί αλλιώ. Τώρα δεν πρέπει να συνδέουμε τη δημοσιονομική στήριξη με την κάλυψη προϋποθέσεων οικονομικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να δυσκολεύσουν τις προσπάθειες των δικαιούχων χωρών προκειμένου να αναπτυχθούν. Όμως, όμως πρέπει να επιμείνουμε ότι ο κύριος στόχος μας είναι η ανάπτυξη, η υποχώρηση της ένδειας, η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας κλπ. Και πιστεύω επίσης, ή τουλάχιστον αυτή είναι η θέση μας, των σοσιαλιστών δηλαδή και δημοκρατών, πρέπει να δώσουμε κίνητρα ώστε οι πόροι που γράφονται στη δημοσιονομική στήριξη να ενισχύουν ε, τα συστήματα βασικών υπηρεσιών. Υγεία, εκπαίδευση, υποδομές, Όλα αυτά δηλαδή που βοηθούν τη χώρα στο σύνολό της και όχι προκειμένου να λυθούν ε, πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε επίσης τον ρόλο που έχουν να παίξουν τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά την απόδοση λογαριασμών. Νομίζω ότι πάντα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίζουμε το ρόλο μας που είναι ο έλεγχος των ε, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επιπλέον να απαιτούμε, να συνεργαζόμαστε, να βοηθάμε την ενίσχυση των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά την απόδοση λογαριασμών. Τέλος, όπως είπε και ο κύριος Γκέρενς, να ενισχύσουμε την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Κοινωνία των πολιτών που και αυτή μπαίνει στα ίδια πλαίσια. Δηλαδή μας ενδιαφέρει η χώρα, οι δομές, οι κοινωνικές δομές. Πρέπει να τις δημιουργήσουμε έτσι ώστε η απόδοση λογαριασμών να ξεπερνάει την αγορά και τις οικονομικές συνθήκες. Όπως είπε και ο κύριος Γκέρενς, και όπως είπε και ο εμπειρογνώμων υπάρχουν τα συν και τα πλην. Υπάρχουν ε, δυνατότητες, αλλοχεύουν και κίνδυνοι. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε στο ιδεώδες μείγμα το καλύτερο ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και να αποφεληθούμε από τις δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Γκέρνς για το έγγραφο εργασία σας. Νομίζω ότι συμφωνούμε με την κριτική σας. Αν και θα το έβλεπα πιο θετικά εγώ, γιατί υπάρχει πολύ δυναμικό. Άλλωστε δεν μπορούμε να εξετάζουμε όλα τα έργα στις χώρες εταίρους. Είναι σημαντικό και για την ιδιοκτησία και για την εταιρική σχέση να υπάρχουν τέτοιου είδους ε, ε, έργα με στήριξη δημοσιονομική. Σημαντικό είναι τώρα να ενισχύσουμε και τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και τον έλεγχο της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων ελέγχου, ελεγκτικά συνέδρια κλπ. για καλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, όχι μόνο προς τους δωρητές και τις ε, παραλήπτριες κυβερνήσεις αλλά και τον ντόπιο πληθυσμό και τους ψηφοφόρους της χώρες εταίρους όπως και ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, βλέπω τους κινδύνους βεβαίως, πρέπει να δούμε πώς θα ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Κίνδυνοι πάντα θα υπάρχουν και ως ένα βαθμό είναι και αποδεκτό αυτό. Είναι οι κίνδυνοι που δεν εξαλείφονται πρέπει να ε, τους δεχτούμε και να τους λαμβάνουμε υπόψη. Κάποιο ρίσκο θα παίρνουμε, αλλά πρέπει οι κίνδυνοι να ελαχιστοποιούνται και η Κομισιόν θα προτείνει και ένα σχέδιο ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Και εμείς θα πρέπει βέβαια να δούμε όλο το δυναμικό που προσφέρει η δημοσιονομική στήριξη στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέρμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δημοσιονομική στήριξη. Σημαίνει ότι στηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών και τα κοινοβούλια προκειμένου να μπορούν να ελέγξουν τι συμβαίνει με τα χρήματα, τι συμβαίνει με τις δαπάνες που κάνει η κυβέρνησή τους. Το να επενδύσουμε στις δυνατότητες αυτές που έχει η κοινωνία των πολιτών και τα κοινοβούλια είναι κάτι που πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Το τονίζω αυτό. Δυστυχώ όμω δεν βλέπω να είναι όντω τέτοια προτεραιότητα και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή. Ε, Πώ επίση. Ε, το ελεκτικό συνέδριο. Ανέφερε κάποια προβλήματα όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη. 35% των πληρωμών που γίνονται για δημοσιονομική στήριξη φαίνεται ότι δεν γίνονται όπως πρέπει. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι το ελεκτικό συνέδριο ζητάει καλύτερο έλεγχο, καλύτερες ε, μεθόδους, καλύτερους ε, δείκτες και αποτελέσματα προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας και το, ελεγκτικό, και το Συμβούλιο, και το Συμβούλιο θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει εδώ το Συμβούλιο, είναι κανείς εδώ από το Συμβούλιο. Συμβούλιο, πουθενά, ναι, όχι, όχι, δεν μπορούν να μου απαντήσουν. Εγώ θα ρωτήσω παρόλα αυτά. Λοιπόν, στα κράτη-μέλη ακούγεται επίσης κριτική από εθνικούς βουλευτές όσον αφορά την δημοσιονομική στήριξη ότι ακριβώς επειδή πολλά πάνε στραβά, ότι εξαφανίζονται χρήματα σε ιδιωτικούς λογαριασμούς κτλ. Στο Συμβούλιο πώς έχει προχωρήσει αυτή η συζήτηση και τι πιθανότητες υπάρχουν όντως να γίνεται κατάχρηση της δημοσιονομικής στήριξης και να πηγαίνουν εξαιτία κακής διακυβέρνησης σε λάθος χέρια. Πολύ θα ήθελα να ξέρω και από την Επιτροπή πώς προχωράει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή έχει το λόγο με τον κύριο Κορέρα Νούνες. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που προσκαλέσατε την Επιτροπή σε αυτή τη συζήτηση και να αποφανθεί για το θέμα αυτό διάβασα την έκθεση του κυρίου Γκέρενς με ιδιαίτερη προσοχή και δεν βλέπω να υπάρχει αρνητική σχέση. Ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις κρίσιμες πτυχές της προσέγγισης της στήριξης των προπολογισμών. Σίγουρα υπάρχουν θετικές πτυχές, όμως ο ίδιος ο συγκητής το αναγνωρίζει. Το να επικεντρωθούμε όμω στι κρίσιμε πτυχέ, στι κρίσιμε διαστάσει, σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τι χρήση βελτίωση. Στον τομέα της βοήθειας η Επιτροπή πάντοτε έχει διαδραματίσει ένα ρόλο καινοτόμο και έχει καταφέρει να προσελκύσει δωρητές γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητηθεί το θέμα της βοήθειας. Αυτό και για την ε, στήριξη των προπολογισμών. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές της δεκαετίας του 90, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των διαφορετικών προγραμμάτων του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου είχε καθοριστικό ρόλο για τη συζήτηση της κατανομής των κονδυλίων. Και θα έρθω στο ερώτημα που έθεσε και ο κύριος Γκέρενς. Ήδη τότε στο επίπεδο του Ταμείου είχε δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της κοινωνικής διάστασης, εκπαίδευση, υγεία. Εκεί ξεκίνησε και η όλη προσπάθειά μας για τη στήριξη των υπολογισμών. Έπειτα είχαμε την ανακοίνωση του 2000 για την στήριξη των υπολογισμών, τη δημοσιονομική στήριξη που έθεσε τα βασικά θεμέλια αυτής της προσέγγισης σε ό,τι αφορά το να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στα αποτελέσματα αλλά και τις αρχές που αργότερα συμπεριλήφθησαν στην ατζέντα των Παρισίων όπως το ownership, η οδικτησία, οι εθνικές ευθύνες, η εναρμόνιση, ο συντονισμός, η καλύτερη ευθυγράμμιση ως προς τις ε, πολιτικές και τη διακυβέρνηση. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. Στα, στο επίπεδο τώρα του πράσινου βιβλίου που έτυχε θετικότατη υποδοχή από όσους το σχολίασαν, Πρέπει να πούμε εδώ ότι η Επιτροπή έπεθε επιτάπητος όλα τα προβλήματα επί των οποίων θα πρέπει να αποφανθούμε στο επίπεδο του Πράσινου Βιβλίου. Υπάρχει ένας κατάλογος προτεραιοτήτων στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Το όλο θέμα της διακυβέρνησης δηλαδή. Εδώ θα πρέπει να εργαστούμε κάποιος πιο σκληρά. Ω τώρα επικεντρωθήκαμε στην οικονομική διακυβέρνηση, τα θέματα που έχουν σχέση με, τα... με τους προπολογισμού, και το μακροοικονομικό πλαίσιο. Πρέπει όμω να καταλάβουμε καλύτερα τη διάρθρωση μεταξύ τη οικονομική διακυβέρνηση και τη πολιτική διακυβέρνηση. Δεδομένη τη πολιτική ευαισθησία του προπολογισμού. Το πεδίο αυτό μελέτης είναι ιδιαίτερα σοβαρό και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Το αναφέρει και η έκθεσή σα. Ένα άλλο μεγάλο πεδίο δράση για μα θα είναι το θέμα των αποτελεσμάτων. Έχουμε προβλέψει δείκτε για τα αποτελέσματα. Οι δείκτε αυτέ συνδέονται με διαδικασίε που είναι πολύ αργές δυστυχώ, είναι βραδίες, έτσι λειτουργεί η ανάπτυξη και είναι πολύ εύκολο είναι μάλλον πολύ δύσκολο να αποτιμήσουμε ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι το χτίσιμο ενός σχολείου, ενός εκπαιδευτικού κέντρου. Μιλάμε για διαδικασίες αργές, βραδίες, ε, που 10-15 χρόνια μετά μπορούν να δώσουν καρπού. Όμως έχουμε κάνει προσπάθειες και ως προς αυτό το θέμα για να αποτιμούμε σωστά τα αποτελέσματα. Για τις ερωτήσεις πάλι που τέθηκαν. Το θέμα του συντονισμού με το Ταμείο, την Τράπεζα και τους άλλους δωρητές. Όπως είπα, η Επιτροπή ανέκαθεν διαδραμάτιζε εδώ σημαντικό ρόλο. Έχουμε ξεκινήσει σημαντικό διάλογο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα με συγκεκριμένα παραδείγματα ανέφερα προηγουμένως τα διευθυντικά προγράμματα, τα παραδείγματα συντονισμού στην πράξη ως προς την στήριξη του υποπολογισμού, τον στατηγικό συντονισμό με τους εταίρους μας και με άλλους δωρητές και με τα κράτη-μέλη. Όπως τα ξέρετε, στα περισσότερα κράτη που προσφέρουν στήριξη στον προπολογισμό, η στήριξη αυτή προσφέρεται από ομάδες δωρητών. μετά από διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με τις κυβερνήσεις. Εδώ είναι καλό βεβαίω να απευθυνόμαστε σε μια και μόνο κυβέρνηση που έχει ένα και μόνο προπολογισμό και μια και μόνο δημοσιονομική πολιτική. Αυτά στο επίπεδο του συντονισμού μα με του άλλου εταίρου. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σχετικά προβλήματα. Πάντως η Επιτροπή είναι σε θέση να οργανώσει διάλογο με τους άλλους εταίρους, προς όφελος βεβαίως των δικαιούχων χωρών. Το όλο ζήτημα των ανταλλαγμάτων για τις χώρες όπου δεν υπάρχει στήριξη στον υπολογισμό. Εδώ έχουμε μια ολόκληρη διαδικασία, μια, ένα ολόκληρο πλωστάσιο ε, στρατηγική που καταρτίζεται και πολύ συγκεκριμένα μέσα. Το γεγονός ότι μια χώρα υποφελείται της δημοσιονομικής βοήθειας δεν σημαίνει ότι λαμβάνει μεγαλύτερη στήριξη από μια χώρα που δεν λαμβάνει τέτοια στήριξη στον προπολογισμό. Αυτό έχει να κάνει με το επίπεδο ανάπτυξη, τον πληθυσμό, την εσωτερική ασφάλεια. Ξέρετε ότι οι χώρες που έχουν χρηστή διαχείριση των ε, δημόσιων οικονομικών τους ε, ένα σωστό μακροοικονομικό πλαίσιο και ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας με καλή διάρθρωση σε συνολικό αλλά και τομεακό επίπεδο προφανώς στηρίζονται στον προπολογισμό τους. Αυτή είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος για αυτές τις χώρες. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπε που δεν στηρίζονται δημοσιονομικώς ποινικοποιούνται. Δηλαδή αντιμετωπίζουν κυρώσει. Εδώ όταν υπάρχει θέμα μη χρηστής διαχείρισης ε, των δημόσιων οικονομικών, όταν υπάρχουν άλλες δυσκολίες, η Επιτροπή αναγκάζεται να βρει και άλλες μεθόδους προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε χώρας. Τους ε, πολλαπλούς δωρητές, την ομάδα δηλαδή ρητών και ούτω καθεξής. Τώρα τι γίνεται με την διακοπή βοήθειας προς μια χώρα. Δώσαμε το παράδειγμα της ακτής του ελεφαντοστού. Πιστεύω ότι ω προ την ιστορία και πάλι η Επιτροπή υπήρξε ανέκαθεν ένα από του πρώτου δωρητέ που ασχολήθηκε με την κατάσταση μια χώρα στην ευρύτερη γεωγραφική τη περιοχή. Την περιφερειακή διάσταση τη διαφορετική βοήθεια δηλαδή. Εδώ λοιπόν ασχολούμαστε με συγκεκριμένε επιπτώσει, το λεγόμενο φαινόμενο spillover, στο σύνολο των εταίρων και συνεργατών σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό ισχύει σε συγκεκριμένες ε, ε, γεωγραφικές ζώνες ε, για χώρες όπως τις λεγόμενες ΕΜΟ, της ΚΟΑΣ και ούτω καθεξής. Η ακτή του ελεφαντοστού του συμμετέχει σε γεωγραφική διαδικασία στο επίπεδο των ΕΜΟΑ και των ΚΟΑΣ και βλέπουμε η συμμετοχή της ακτής ελεφαντοστού τι επίδραση έχει στους υπολείπους, τη λήψη των αποφάσεων. Έτσι καθορίζουμε και εμείς πώς θα δώσουμε τη βοήθειά μας. Εάν υπάρχουν λοιπόν θεσμικές διαδικασίες βάσει του άρθρου 96 που περιγράφονται με μεγάλη σαφήνεια, βλέπουμε τι γίνεται στις επιμέρους περιοχές. Ναι λοιπόν αυτή είναι μια μέρημνα που την έχουμε διαρκώς. Ο ρόλος των χρόνων αυτών σε ε, περιφερειακό επίπεδο. Και για το τελευταίο σας ερώτημα επειδή είπα ότι η στήριξη δημοσιονομική είναι ο καλύτερος τρόπος να αναπτυχθεί μια χώρα εσωτερικός, εμβογενός. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, υπάρχουν και άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η καλή οικονομική διακυβέρνηση κατά πρώτον. Εάν τα κριτήρια αυτά πληρούνται, η στήριξη του για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά για να γίνει και ενδογενής, εσωτερική δηλαδή αυτή η ανάπτυξη. Έτσι, εντασσόμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό που είναι προς όφελος και των ίδιων των χωρών, αλλά και εναρμόνισης και συνεργασίες με άλλους δωρητέ και εταίρους. Για να ολοκληρώσω λοιπόν. Μιλήσαμε και για το ελεκτικό συνέδριο. Βεβαίω το ελεκτικό συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του προπολογισμού, για την συμμόρφωση και το σεβασμό των κανόνων. Εσείς ως Ευρωκοινοβούλιο είσαστε ένα άλλο θεσμικό όργανο δημοσιονομικού ελέγχου. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις που ήδη εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του, αλλά κυρίως δύο είναι οι βασικές διαστάσεις επί των οποίων θα πρέπει να εργαστούμε. Πρώτη, η διακυβέρνηση και έπειτα τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την δυναμική μας προσέγγιση, μιλώ για την οικονομική διακυβέρνηση, μιλήσατε για τα δημοσιονομικά και το μακρονομικό επίπεδο. Εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτής της δυναμικής προσέγγισης, όμως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκροτημένοι στην ανάλυση μας. Δηλαδή από τη μια περίοδο στην άλλη να βλέπουμε τι βελτιώσεις έχουν επιτευχθεί τι πρόοδο υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο. Από αυτού συμφωνούμε απολύτω με τι θέσει του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα πρέπει να Είμαστε πολύ πιο σαφείς ότι η ανάλυση θα ακολουθήσουμε ως προς την οικονομική διακυβέρνηση. Ως προς τα αποτελέσματα, το συνέδριο εντόπισε κάποιες ελλείψεις και κενά που θα πρέπει να καλυφθούν, όμως θα πρέπει να προσέξουμε κάτι άλλο που είναι σημαντικό όταν μιλούμε για αποτελέσματα. Από τη μια έχουμε τη στήριξη τη δημοσιονομική και από την άλλη τους δείκτες. Και ποια είναι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να αποφύγουμε τις σχέσεις αιτίου αιτιατού. Δεν σημαίνει ότι η στήριξη της Επιτροπής είναι υπεύθυνη για όλα τα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Συμμετέχουμε σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, όπου υπάρχει και η πολιτική της κάθε χώρας, υπάρχει η παρουσία της Επιτροπής, αλλά και άλλων εταίρων. Ειδού Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν ξέχασα τίποτα. Ως προς τις ερωτήσεις που τέθηκαν, ελπίζω ότι σας κάλυψα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μόρα Σαν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Εμείς συμμετέχουμε και συμφωνούμε. Όμως εμένουμε στην θέση μας για το ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε κάπως πιο ανοιχτά τις τρεις πτυχές της επιλεξιμότητας για να δοθεί η δημοσιονομική στήριξη. Δεν έχει γίνει συζήτηση για το τρόπο που έχει εφαρμοστεί ε, έχουν εφαρμοστεί αυτά τα τρία κριτήρια στο παρελθόν και αν θα έπρεπε κάτι να αλλάξει. Εμείς οι πυρογνώμονες έχουμε ασχοληθεί με αυτό και έχουμε καταλήξει στην απόψή μας όπως επίσης και το θέμα του πώς επηρεάζουν τα συστήματα λογοδοσίας από τις χώρες δωρητές που είναι διαφορετικό. Υπάρχει διαφοροποίηση στην διεθνή συνεργασία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρε που είναι πολύ επιφυλακτικές όσον αφορά την διμερή συνεργασία. Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν τη δημοσιονομική στήριξη για να προβάλλουν περισσότερο τα συμφέροντά τους. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφοροποίηση. Και πολλές χώρες δικαιούχοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με τα διαφορετικά αυτά συστήματα Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι πάντα αρνητικό. Αλλά λέμε ότι θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση και στην πράσινη βίβλο για την εμπειρία που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα και πώς εκτιμάει και αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εμπειρία αυτή όταν υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια σε εθνικό επίπεδο και από πλευράς των ε, δωρητών όταν είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες, δηλαδή απόδοσης λογαριασμών, πώς, ε, όταν είναι διαφορετικά τα κριτήρια, πώς αυτό επηρεάζει την όλη κατάσταση. Όπως λέει και ο κύριος Κορέα Νούνιες, ανοιχτά έχουν μπει σε συζήτηση τα διάφορα θέματα του μέσου αυτού. Σίγουρα η πράσινη βίβλος είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Απλώς θέλουμε εμείς κάποια σημεία να είχαν αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο μέσα στην πράσινη αυτή βίβλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκέρενς τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από τη συζήτηση αυτή, και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο, όλους και εσάς, τον εμπειρογνώμων, αλλά και όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να πω ότι η συζήτηση με ενθαρρύνει, γιατί βλέπω ότι συγκλίνουν οι απόψεις μας τελικά. Οι πιο επικριτικές μου παρατηρήσεις είναι παρατηρήσεις με τις οποίες συμφωνούν και οι υπόλοιποι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην περιφερειακή διάσταση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, η Κομισιόν είναι ο πιο σημαντικός ε, χορηγός βοήθειας η περιφερειακή διάσταση λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν ε, μέσα, άλλα πέρα από αυτό που συζητάμε εδώ, που εθαρρύνουν την περιφερειακή διάσταση. Και σημειώνω αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει εφόσον μια χώρα δικαιούχος δεν έχει το κεκτημένο που θα έπρεπε. Από ό,τι κατάλαβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να διορθώσει τις αδυναμίες. Δεύτερη τυχή, ownership, ποιος δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο είδους ανάληψη ευθύνης, δεν υπάρχει και ανάπτυξη. Αυτό είναι το βασικό θεμέλιο, η βασική αρχή που διέπει όλη μας την προσπάθεια. Αυτό ισχύει και για την Ευρώπη. Το κοινωνικό μοντέλο των σκανδονοβικών χωρών είναι ακριβώ ένα μοντέλο που βασίζεται στην ανέλυψη ευθύνη και το οικονομικό μοντέλο τη Μεγάλη Βρετανία το ίδιο. Ε, εάν όμω ε, ανταλλαχθούν τα δύο μεταξύ του, δεν θα λειτουργούν. Θα πρέπει λοιπόν για να προσαρμοστεί κανεί ένα σύστημα να έχει χρόνο στη διάθεσή του. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και επαρκή κατανόηση από τι ε, χώρε εταίρου μα στο Νότο. Τώρα, ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και την αποτίμηση, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, θα πρέπει στους όρους αναφοράς, για να τους πούμε έτσι, τα κριτήρια θα πρέπει ήδη να περιέχουν τους όρους αναφοράς της αξιολόγησης. Θα πρέπει δηλαδή από την έναρξη της στήριξης της δημοσιονομικής να γνωρίζει κανείς ποια είναι τα κριτήρια, τα στοιχεία βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί στη συνέχεια. Πρόκειται για μια διαδικασία διαρκείας. Είναι νομίζω αυτονόητο σχεδόν, αλλά κάποιες φορές κινδυνεύουμε να το ξεχνούμε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένα μόνιμο αντανακλαστικό μας για κάθε πολιτική συνεργασία αναπτυξιακής δεν μπορούμε εκ των υστέρων να επινοούμε τα κριτήρια, θα πρέπει να έχουν επινοηθεί ευθύ εξ αρχή. Οπότε ο καθένα ξέρει ακριβώ τι να περιμένει και να ξέρει και βάσει ποιων κριτηρίων θα στηριχθεί. Τρίτη πτυχή. Τέταρτη μάλλον. Δεν μπορώ παρά να κάνω μία παρατηρήση για αυτό που θα ονόμαζα αμφίσιμη στάση των κρατών μας. Από τη μια όλοι δέχονται τη δημοσιονομική στήριξη, και αυτό βάσει και τις εντολής που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τα κράτη στο εσωτερικό τους, από μόνα τους μάλλον, επιφυλάσσονται και δεν ε, κάνουν τέτοια ίδια βοήθεια, διστάζουν. Αυτό ενέχει από μόνο το ένα κίνδυνο και είναι ένα βασικό στοιχείο, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε το ρίσκο. Μια πολιτική όμως χωρίς ένα βαθμό κινδύνου. Εφόσον μιλάμε για ανάπτυξη και εφόσον υπάρχουν εξελίξεις καθημερινά, κάθε μέρα μαθαίνουμε νέα στοιχεία. Αυτό δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη μία αποδοχή μιας ε, βασικής έννοιας, ενός βασικού βαθμού κινδύνου. Θα μας έκανε κάτι τέτοιο, εάν γινόταν αποδεκτό, να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να έχουμε νομίζω το θάρρος και την τόλμη να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Κάθε πολιτική, είτε είναι εκπαιδευτική, είτε οικονομική, είτε περιφερειακής βοήθειας, ενέχει και ένα βαθμό απολειών. Πρέπει να είμαστε τολμηροί και να μπορούμε να το πούμε. Τώρα, εάν στις αξιολογήσεις μας δεν αποκαλύπτουμε αυτό το μικρό βαθμό απολειών, δεν είμαστε εντάξει. Εκεί θα αρχίσει κανείς να διερωτάται αν αξίζει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου. Ας είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι και ας φροντίσουμε οι απώλειες να είναι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο υποφερτό. Γιατί αλλιώ δεν έχει νόημα το σύστημα ανείχνευση των ε, πολιών, αλλά και αν δεν τι αποκαλύπτουμε πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε. Σαν να μην υπήρχε. Α είμαστε λοιπόν τολμηροί και να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Για τα 50 δις δολάρια, μάλλον ευρώ που δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση, 5% στα γενικές δαπάνες σπαταλώνται, διασπαθίζονται, χάνονται. Τέλο πάντων δεν εξυπηρέτησαν το σκοπό για τον οποίο αρχικά είχαν αποδοθεί. Αυτό πρέπει να έχουμε τον τόλμη να μπορούμε να το πούμε. Αλλιώ δεν θα έχουμε ποτέ αυτή την ε, αποδοχή του κινδύνου και δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και ένα θετικό σχόλιο, το έγγραφο, όπω είπα και εν είδη εισαγωγή, κυρίω αφήνει ανοιχτά ερωτήματα εκφράζει ανησυχίες Παρουσίαση του εμπειρογνώμονά μας, επιβεβαίωσε τη στάση μας. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν και κίνδυνοι και θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουμε την όλη κατάσταση. Το δυναμικό που έχει αναπτυξιακή βοήθεια νομίζω είναι πολύ σημαντικότερο το άλλο από του κινδύνου. Αρκεί να, γίνει, να μπορεί κανεί να αποδέχεται του κανόνε και να είναι υπεύθυνο στη στάση του. Εδώ είμαστε στην αρχή του όλου επίπονου αυτού έργου. Δεν θέλω στα εισαγωγικά μου σχόλια να ξεπεράσω αυτούς του ε, περιορισμένου τομεί. Θα περάσουμε σε μια νέα φάση συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ευχαριστώ ιδιαίτερω. Νομίζω θα συνεργαστούμε μια χαρά, έτσι είναι εφικτό. Κοιτάξτε. Εντάξει, όπως μου το λες και εσύ, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα συσχετισμό μεταξύ της ε, δημοσιονομικής στήριξης και των κατεξουσιοδότηση πράξεων στο στατηγικό έγγραφο που θα ετοιμάσετε. Υπάρχουν κι άλλα που κυκλοφορούν μέσα από την δημοσιονομική στήριξη. Εμεί εδώ ω βουλευτέ, έχουμε το δικαίωμα να διερωτώμεθα εάν είναι το καλύτερο αυτό μέσο ώστε να ανταποκριθούμε στους τελικού τελικούς στόχους που έχουμε θέσει για στήριξη των ε, πλέον φτωχών, για στήριξη των παραγωγών, ε, για την κάλυψη των περιβαλλοντικών μας μεριμνών. Τρία σημεία στα οποία επιμείναμε στα πλαίσια του γράφου μας. Μη μας στερείτε την εξουσία συμμετοχή που διαθέτουμε στου τομείς αυτούς. Εκεί θα είχαμε μία πίσχναση της πολιτικής ε, της των προσπαθειών μας. Αυτά ήταν τα σχόλια μου. Ε, εάν φάνηκα και λίγο κακός, αυτό έγινε γιατί μέχρι τώρα η Επιτροπή ήταν σχετικός καλή μαζί μας. Ουσιαστικά προσπαθώ να πω στην Επιτροπή ότι δεν είμαστε εδώ ένα σύλλογο ε, γέσμεν. Ευχαριστούμε, θα διακόψουμε τώρα τη συνεδρίασή μας. Να θυμάστε ότι έχουμε ανταλλαγή απόψεων σήμερα στις 3 και τέταρτο, σε κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην αίθουσα 2Q2 ε, για το θέμα της ακτής του ελεφαντοστού. Και έπειτα θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα εδώ.